Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Είναι ήδη 9 και 5. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Σας είπα χθε ότι θέλω να ξεκινήσουμε γέρο σήμερα και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί έχουμε πολλά σημεία στη μερίσια διάταξη. Ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να κάνουμε σήμερα είναι να καλύψουμε όλες αυτές τις ψηφοφορίες. Έξι εκθέσεις συνολικά πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα. Ελπίζω ότι θα κινηθεί ομαλά η ψηφοφορία. Είναι η πρώτη φορά που προεδρεύω επίσημα στη συνεδρίαση αυτή και θα προσπαθήσω να καλύψω στο δυνατόν γρηγορότερα αυτές τις ψηφοφορίες. Λοιπόν, αρχίζουμε αμέσω με την πρώτη έκθεση. Σίλβια Κώστα. Για την έκθεση υλοποίηση εκτέλεση του Creative Europe. Δεν ξέρω αν θέλει να πει τίποτα η συγγήτρια. Όχι. Να σας πω μόνο ότι θέλω να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις συγητές και προφανώς τους policy advisors καθώς επίσης και την γραμματεία για την καταπληκτική συνεργασία που είχαμε και να ευχαριστήσω επίσης και τη συνάδελφο Τζίτζος από τη γραμματεία. Ελπίζω ότι ε, θα κινηθεί ομαλά η ψηφοφορία αυτή και ότι θα μας βρει τελικά όλους σύμφωνους. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, περνούμε αμέσω στη ψηφοφορία. Συμβαστική 1. Ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Στην επόμενη σελίδα η 1 του προϋπολογισμού υπέρ. Budget 1. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Οι δύο της Επιτροπής Προβολογισμών υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία του δεύτερα ψήφι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 88 και 89 που είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. Τροπολογία με 90 υπέρ. Κατά. Ξανά, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η τροπολογία 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε τώρα στην τροπολογία 98 και 99 μαζί υπέρ. Είναι μας εξα... Κατά. Αποχές νομίζω ότι έχει απορριφθεί. Η τροπολογία 100. Ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 104 και 105 μαζί ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται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 118 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 124 επε κατά αποχές απορρίπτεται 125 επέ κατά αποχές εγκρίνεται 126 επέ κατά αποχές απορρίπτεται 127 επέ κατά αποχές απορρίπτεται 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 130 και 131 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 133 γιατί έχει καταπέσει 132 133 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά απόχες εγκρίνεται. Πάμε τώρα στα 142 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. 143 υπέρ κατά αποχές παρακαλώ να το τσεκάρουμε γιατί δεν βλέπω τι γίνεται Αρχίζει ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρα. Έχουμε έναν υπεράριθμο από το ΕΛΚ που ψηφίζει. Einer, Κάντε μια καρτούλα. Πέρασε. 13-12. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Αυτά είναι. 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 145 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 146 υπέρ κατά κατά αποχές εγκρίνεται 147 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 148 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 149 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται 150 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται 151 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται 152 υπέρ κατά αποχές για να το ελέγξουμε παρακαλώ αυτό αρχίζει η ψηφοφορία ψηφίσετε όλοι πέρας Angenommen. Εγκρίνεται. 153 ήταν αυτή. 153 ψηφίζουμε τώρα μάλλον υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δηλαδή απορρίπτεται, διορθώνει η Πρόεδρος. 154 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 157 έχει αποσυρθεί όπως και 158 εδώ έχουμε μια προφορική τροπολογία λέει της εισηγήτριας ψηφιπέ κατά αποχές εγκρίνεται 160 ψηφιπέ κατά Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην 167. 167. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 168 Υπέ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 169 υπέρ. Όχι καταπίπτει φωνές. Α, ναι, ζητώ συγγνώμη λέει η πρόεδρο. Συμβαστική 8. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην 174. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 175 υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται 177 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται 178 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται Πάμε στην 182 μέσος υπέρ κατά απόχες απορρίπτεται 183 υπέρ κατά αποχές λοιπόν ξανά υπέρ κατά Εκατόν υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται σαφέστατα. 184 υπέρ. Α, όχι, έχει καταπέσει. 185, ζητώ συγγνώμη, λέει πρόεδρος, 185 υπέρ. Κατά, άποχε. απορρίπτεται. 186 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 187 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 188 υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι έχει απορριφθεί. 192 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 193 υπέρ. Κατά. Με αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 3 του προπολογισμού υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 199 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε τώρα συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 5 της Επιτροπής Προπολογισμών στην επόμενη σελίδα ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 216 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 217 με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 218 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 219 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 220 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 221 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. 222 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 223 και 224 μαζί είναι μας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 225 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 226 υπέρ. Α, όχι, σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτον υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι πάρα πολύ σαφές. Ας το ελέγξουμε παρακαλώ. Αρχίζει η ψηφοφορία. Geschlossen. Πέρασε abgelehnt. Das Απερίφθη. Α, και σαφέστατα μάλιστα. μάλιστα. Λοιπόν, 227 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 και 17 μαζί όχι, καταπίπτουν και μαζί και 18, 21 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 22 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 23 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 24-25 μαζί, ταυτόσιμες, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται, 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές ας το λέξουμε για καλό και για κακό αρχίζει η ψηφοφορία Πέρας. 14-13 εγκρίνεται. 34. Dafür. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ich Και αυτό χρειάζεται παλήθευση, παρακαλώ. Η Abstimmung ist eröffnet. Έχει την ψηφοφορία. Πέρα. Α, όχι, σαφέστατα εγκρίνεται. Δεν ψηφίζεται. Λοιπόν, 38 είπε, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 40 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 είπε, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 είπε, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Όχι, καταπίπτει. Ε, 43 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά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 Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά δεν είμαι βέβαια. Για να το ελέγξουμε, παρακαλώ, αρχίζει η ψηφοφορία. Geschlossen. Πέρασε. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Απόχε. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. απόχέ, Απορρίπτεται. 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, συμβαστική το 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε αμέσως στην 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία είναι υπέρ κατά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι δύο υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται η 3 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται η 4 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 5 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται η 6 έχει αποσυρθεί 7 και 8 μαζί είπε, κατά αποχές εγκρίνονται 9, 10 και 11 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι έχει εγκριθεί θέλουμε να το ελέγξουμε πάμε αρχής προφορία Πέρας. Ναι, ναι, είχε εγκριθεί. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η ε, αιτιολογική αναφορά citation του προεβολογισμού ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα. Geschlossen. Ε, Εγκρίθηκε 24 ε, ψήφοι υπέρ, καμία κατά, 4 αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Κώστα και σκιώδης συγγητές για τη δουλειά σας και σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάει πρώτη. Προχωρούμε. Είναι για την ε, έκθεση υλοποίησης ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ευρώπης για τους πολίτες. Η συζήτρια ήταν η κυρία Χιμένεθ Μπαρμπάτ. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε τίποτα. Τίποτα, όχι. Απλώς θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεισέφεραν για την έκθεση αυτή και ελπίζω να ε, έρθει σε αίσιο Είναι πάρα πολύ σημαντική έκθεση για προγράμματα που βοηθούν στη συνοχή και στη συνεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ και σας για τη δουλειά σας και τους και σας και πάμε μέσω στην ψηφοφορία. Έχουμε την τροπολογία 53 που δεν μπορούμε να την ψηφίσουμε γιατί είναι απαράδεκτη και πάμε στην τροπολογία 54. Ψηφίπερ. Κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 ε, ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, ε, ένα το προπολογισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ή 60, 61 και 63 ομού. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Ή 62 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. 64 υπέρ. Κατά αποχές απορρίψετε 65 υπέρ κατά αποχές απορρίψετε 66 και 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές. Αυτό θέλει έλεγχο. Πάμε λοιπόν να αρχίσει η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη σαφέστατα. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αύκο 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι, απορρίπτεται, η πρόεδρος. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίψετε 76 υπέρ κατά αποχές απορρίψετε 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές απορρίψετε 80 υπέρ κατά αποχές απορρίψετε 81 υπέρ κατά αποχές. Ας το ελέγξουμε λοιπόν. Αρχίζει η ψηφοφορία στην 81. Πέρας. Απορρίπτεται. 11-13. 82. Ψηφί υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. 84 υπέρ κατά αποχές 84 84 ψηφί κατά αποχές έλεγχος άρχεται ψηφοφορία geschlossen πέρας das ist angenommen εγκρίνεται 85 υπέρ. Όχι, ζητάει συγγνώμη, πρόεδρος 86 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά άποχέ εγκρίνεται. 89 και 90. Α, και 91 και 92. Υπέρ. Κατά. απόχέ, αποχές. Απορρίπτεται 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω και... Die 95. Dafür. Dagegen. Υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 95 ήταν αυτή, 94 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 96 είπε κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 4 είπε κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και πάμε τώρα στην 103. Ψηφί υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 104 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 4 του προβολισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 105 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται. 106 είπε, κατά αποχές Απορρίπτεται. 107. Έχει αποσυρθεί. 108. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 109. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 110. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αύκο 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αύκο 7. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αύκο 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αύκο 9 έλεγχο. Καλώς να το ελέγξουμε. Αρχίζει ψηφοφορία για την ΑΦΚΟ 8. Πέρασε. Σαφέστατα εγκρίθηκε. ΑΦΚΟ 9. Ψηφιπέ κατά αποχές απορρίπτεται 111 ψηφί π. κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αυκό 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην 121 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 123 είπε κατά αποχές απορρίπτεται. 6 ε, του προπολογισμού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 124 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. 125 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. Δηλαδή απορρίπτεται, διορθώνει πρόεδρος. 126 υπέρ κατά απόχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά άποχέ εγκρίνεται. 133 τώρα, γυρνάμε σελίδα. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τελειώνει τώρα. ψηφία απορρίπτεται. 135 ψήφοι υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 149 υπέρ κατά αποχές έλεγχος στην 149 πέρας εγκρίθηκε δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά τα ψηφίζετε 150 είπε. κατά αποχές απορρίφτεται 151 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίψετε. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 154 υπέρ. Και 55, 155 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ. Καλά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Απερίφθη. Ζητώ συγγνώμη, λέει 158 υπέρ κατά αποχές ενδιέται. Η προφορική τροπολογία 2 στην ΑΦΚΟ 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. προφορική τροπολογία 1 στην 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 160 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Και πάμε στην τροπολογία 23 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται αύκο 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 26 ψηφιπε, κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ, κατά, αποχές έλεγχο χρειάζεται νομίζω αυτό. Στην 32 είμαστε. Πέρασε. Τι γίνεται με τα χέρια σας. Λοιπόν, απερίφθη, σαφέστατα. 33, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 34, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπε κατά, αποχές, απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. συγγνώμη. 48 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 49 ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές απορρίψετε, 51 υπέρ, κατά, αποχές απορρίψετε. Die 52 dafür. 52 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα έχουμε και κάτι γνωμοδοτήσεις. Αύκο και budget, αλλά τα έχουμε ψηφίσει ή έχουν καλυφθεί από άλλες τροπολογίες και πάμε στην τελική ψηφοφορία η οποία τροπολογιες και παμε στη τελικη ψηφοφορια που Πέρασε. 24 υπέρ, 5 κατά, χωρίς αποχές, εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια, κυρία Συγγήτρια. Και σε ελπίσουμε να ευδοκιμήσει η Ευρώπη για τους πολίτες και μάλιστα γρήγορα. Επόμενη ψηφοφορία, παριθμόν 3. Για το γεωγραφικό αποκλεισμό, λεγόμενο και geo-blocking. Η συγκίτρια ήταν η κυρία Κομοδίνη. Θέλετε να πείτε τίποτα? Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω απλώ όλου του κοιόδη ηγητέ και όλου του συμβούλου μα που μα βοήθησαν πάρα πολύ για την επεξεργασία αυτή τη πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε με στην ψηφοφορία. 93 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 97 και 24 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 102 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 103 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 είπε κατά αποχές απορρίπτεται 31 ε, παρακαλώ υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι έχει απορριφθεί αλλά θέλω να το ελέγξουμε παρακαλώ αρχίζει η ψηφοφορία στην τροπολογία 31 Πέρας. Απερίφθηνε. 115 υπέρ. Κατά. Ε, αποχές απορρίπτεται. 117 υπέρ. Κατά. Α, 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 119 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 120 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 123 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογή παρθών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 36 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ή 42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές απόρριψεται 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 49 ναι. υπέρ κατά απόχέ απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία παριθμών λοιπόν, 6 τώρα ψήφι υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές απόρριψη 64 υπέρ κατά αποχές απόρριψη 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 είπε. κατά αποχές νομίζω ότι θέλει έλεγχο αρχίζει η ψηφοφορία για την τροπολογία 69 Πέρασε. Ισοψηφία, άρα απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 74 είπε, κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 είπε, κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές Παρακαλώ να το τσεκάρουμε. Αρχίζει η ψηφοφορία, είναι στην τροπολογία 17. Geschlossen. Απερίφθη. 79 ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Πού πάμε τώρα. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, η 91 υπέρ, κατά άποχες, απορρίπτεται, η 92 υπέρ, κατά άποχες, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Αρχίζει τώρα, παρακαλώ. Geschlossen. Πέρασε. 21 ψήφοι υπέρ, μία κατά, 5 σε Συγχαρητήρια, κυρία Κομοντίνη. Λοιπόν, έχουμε άλλες τρεις. Έκθεση του κυρίου Τζαμπάρσκι τώρα για την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Δεν ξέρω αν θέλει να πει τίποτα ο εισηγητής. Δεν θέλει. Καλώς. Πάμε στην ψηφοφορία λοιπόν. Κατευθείαν. Συμβαστική 1 είπε. Κατά. Αποχές εντυρίνεται. Τροπολογία 7 είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές αυτό μάλλον θέλει έλεγχο παρακαλώ τροπολογία 10 αρχίζει η ψηφοφορία πέρασε απερίφθη Συμβαστική 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 15 είπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Τι 12. Εδώ είστε. Α, καλά. Γλίστρισα. 17 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος παρακαλώ στις 17 αρχές ψηφοφορία πέρας εγκριθήκε 16-10 τροπολογία 18 σε δύο τμήματα τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε μέσω στην 34 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος παρακαλώ. Αρχίζει ψηφοφορία. Geschlossen. Πέρας. 16-10 ε, εγκρίνεται. Εγκρίνεται 16-10. 36 πέρα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ κατά αποχές παρακαλώ να το ελέγξουμε αυτό Geschlossen. Τέλος. Απερίφθη. 10 υπέρ, 15 κατά. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πώς θα ξεπετάμε. Τελική ψηφοφορία. Αρχίζει τώρα. Πέρας. Τώρα. Ομόφωνα. 26 υπέρ, χωρίς αποχές και χωρίς αντίθετες ψήφου. Συγχαρητήρια κύριε Τζαμπάτσκι. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Πρώτη τελευταία ψηφοφορία για σήμερα για την απαλλαγή για τον προπολογισμό του 2015. Η συγκεκριά ήταν η Σίλβια Κώστα. Θες να πεις τίποτα, Σίλβια? Ε, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω απλώς για... Μάλλον να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία και τη γραμματεία. Τελικώς ε, προσπαθήσαμε να είμαστε πολύ συγκεκριμένη και ακριβή να σας ζητήσαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφίζουμε λοιπόν τροπολογία 1, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, η 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, η 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, πέντε υπέρ,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 Πέρας. Εγκρίνεται 21 ψήφι υπέρ, 1 κατά και 4 αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Κώστα. Και πάμε τώρα στην τελευταία μας ψηφοφορία για σήμερα. Εντάξει, αρκετά ψηφίσαμε για σήμερα. Είναι λέει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και ο συντονισμό οικονομική πολιτική. Η συγγήτρια κυρία Τζούλι Γουόρντ. Θες να πει τίποτα Τζούλι? Πολύ σύντομα, Πρόεδρε, γιατί, όπως είπατε, αρκετή ώρα ψηφίζουμε. Εδώ προσπαθούμε να εγγυηθούμε τα δικαιώματα των παιδιών, γιατί το εγγυητικό μέσο είναι τμήμα αυτής της βιάση και αρκετοί συνάδελφοι έχουν συνεργαστεί μαζί μου για τα δικαιώματα των παιδιών στις ομάδες. Ήθελα απλώς να κατανοήσουν οι συνάδελφοι ότι αυτό ψηφίζουμε σήμερα για τα παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αμέσως ψηφίζουμε. Τροπολογία 1, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές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 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα που πάμε Σε 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι έχει απορριφθεί αλλά ας το καλύτερα 47 με μικρή διαφορά ενέντε.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 τελειώνει. Εγκρίνεται η έκθεση με 22 ψήφου υπέρ, 4 κατά χωρί αποχέ. Συγχαρητήρια κυρία Γουόρτ. Πάει και αυτό. Τα καταφέραμε. Μαμούθ η ψηφοφορία αυτή. Καλά τα πήγαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συγκέντρωση και τη συνεργασία. Και να με συμπαθάτε πρώτη φορά προεδρεύω σε ψηφοφορία.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 Λοιπόν, συνεχίζουμε αμέσω. δεν έχει διαλύματα και τέτοια. Απλώς περιμένουμε, περιμένουμε να έρθει η Μαλτέζικη Προεδρία, οι δύο υπουργοί που περιμένουν, περίμεναν να τελειώσουν την ψηφοφορία μα και θα συνεχίσουμε αμέσω μετά.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 Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ich würde gerne mit unserer ε, θα ήθελα να συνεχίσουμε με ιδιαίτερη χαρά και τιμή καλωσορίζω σήμερα τους εκπροσώπους της ε, Βαλτέζικης Προεδρίας και μάλιστα τους Υπουργούς Μπάρτολο και Μπονίτσι στην Επιτροπή μας. Χαίρομαι πάρα πολύ που ε, ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή μας για να μας παρουσιάσετε τις προτεραιότητες της Προεδρίας της χώρας σας στους ε, τομείς ε, που ενδιαφέρουν την Επιτροπή μας και είναι της δικής μας αρμοδιότητας. Ξέρω τι σημαίνει για μια μικρή χώρα να προεδρεύει στο Συμβούλιο. Σας παρακαλώ κάντε λίγο Έλεγα λοιπόν ότι είναι μεγάλη πρόκληση για μια μικρή χώρα όπως τη Μάλτα να αναλαμβάνει ε, την Προεδρία των 28 ακόμα κρατών μελών, αλλά ε, είμαι σίγουρη ότι θα αξιοποιήσετε πάρα πολύ καλά το εξάμεινο αυτό που σας αναλογεί, έτσι ώστε να προωθήσετε και θέματα ε, που είναι ειδικού ενδιαφέροντος για μας και να πάτε λίγο, παραπέρα, λίγο παρακάτω την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας δώσω το λόγο για 10 λεπτά στον καθένα να μας παρουσιάσετε τις προτεραιότητές σας και στη συνέχεια θα περάσουμε στη συζήτηση. Χρόνο έχουμε μέχρι τις 11.30. Νομίζω ότι θα είναι καλή συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στον Υπουργό κύριο Μπαρτόλο πρώτα, που είναι αρμόδιος για θέματα παιδείας και απασχόλησης. Ε, είναι θέμα αυτό πάρα πολύ σημαντικό για την Επιτροπή μας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Υπουργέ. Καλώς ορίσατε και πάλι στην Επιτροπή μας. Good morning. Good morning. Καλημέρα. Καλημέρα Πρόεδρε, καλημέρα αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι. Να σας ευχηθώ και καλή συνέχεια και καλή επιτυχία για τη δουλειά σας εδώ ως Πρόεδρος και να ευχαριστήσω και την κυρία Κώστα για τη δουλειά που έκανε, λέει ο μιλητής στα Ιταλικά, την προηγούμενη περίοδο. Τώρα θα συνεχίσω στα Μαλτέζικα. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ότι αυτή εδώ η στιγμή είναι πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δύσκολη η καιρή. Ε, εκφράζονται αμφιβολίες ε, σχετικά, για το λόγο, σχετικά με το λόγο ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμα. Ε, και κάποιοι θέλουν να φορτώσουν τις ευθύνες των όσων συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλησιάζοντας και την 60η επέτειο της ίδρυσης, πρέπει να δείξουμε ότι αντιθέτως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κομμάτι της λύσεως, της διεξόδου από τα όσα αντιμετωπίζουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση <clears throat> που αντιμετωπίζουμε είναι ακριβώς να μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με πιο άμεσο τρόπο με τους πολίτες γιατί αυτοί που προσπαθούν να βλάψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάρα πολύ καλοί σε θέματα επικοινωνίας. Δεν πρέπει λοιπόν να τους επιτρέψουμε να μας υπερφαλαγγίσουν στην επικοινωνία αυτή. Θα πρέπει να δείξουμε στους πολίτες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για τα θέματα που απασχολούν καθημερινά τους πολίτες και συζητούν καθημερινά. Ότι μπορούμε να υπηρετήσουμε τους πολίτες σε διάφορα πεδία, στα θέματα της νεολαίας, του πολιτισμού, του αθλητισμού μεταξύ άλλων. Πρέπει να τους δείξουμε πάντως <clears throat> ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητη. Και να σας ε, πω και δύο λόγια ε, για το τι σκοπεύουμε να κάνουμε στο εξάμεινο της Προεδρίας μας ε, στα θέματα ακριβώς αυτά παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού. Στην παιδεία οι βασικές προτεραιότητες είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα στα οποία κάποιοι αισθάνονται ότι τους έχουμε ξεχάσει. Αυτά είναι τα θέματα της ανεργίας, όχι μόνο από την ασθενή οικονομική μεγέθυνση, αλλά και την αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων. Έχουμε θέσεις απασχόλησης διαθέσιμες, αλλά Πολλοί άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι να τις καλύψουν γιατί δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Η θεματική προτεραιότητα λοιπόν της ε, ανώτατης παιδείας για όλους της Προεδρίας είναι απολύτως επίκαιρη διότι το 11% των νέων εγκαταλείπουν το σχολείο νωρίτερα το 70% δεν συμμετέχει σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης ε, προς την επαγγελματική απασχόληση. Έχουμε υψηλά ποσοστά χαμηλών δεξιοτήτων και πολύ σημαντικό ποσοστό 44% που αισθάνεται ότι δεν έχει την ευκαιρία με τις δεξιότητες και τα προσόντα που έχει στην αγορά εργασίας. Έχουμε λοιπόν και το θεματολόγιο των δεξιοτήτων και τη δέσμευσή μας ε, στην διαβίου μάθηση. Κάτι πρέπει να επικαιροποιούμε και θα επικαιροποιήσουμε και με το νέο πλαίσιο ακριβώς της διαβίου μαθήσεως. Και που είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για τους ανέργους, αλλά για όλους, γιατί γνωρίζουμε ότι σήμερα ότι πρέπει συνεχώς να ενημερώνουμε τις δεξιότητές μας δυναμικά. Και στην ενότητα παιδεία για όλους προσπαθούμε να υπογραμμίσουμε την διαφορετικότητα και την ένταξη και μιλούμε για ένα ευρύτατο φάσμα ανθρώπων και τους μετανάστες και τα παιδιά των μεταναστών και τους ανθρώπους με αναπηρία και τους ανθρώπους με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Διαφορετικότητα λοιπόν όπως την κατανοεί κανείς με την ευρεία τη δυνατή ερμηνεία. Και ένταξη συμπερίληψη όχι φασών πρέπει να έχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες πολλών διαφορετικών ανθρώπων. Γιατί για πάρα πολλά χρόνια τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη ήταν συστηματοποιημένα. Περιμέναμε λοιπόν όλοι οι άνθρωποι να χωρέσουν στο σύστημα έτσι όπως αυτό είχε σχεδιαστεί. Πρέπει να καλύψουμε διαφορετικές ανάγκες πλέον. Και αυτή την αρχή θα την προωθήσουμε υπό την Προεδρία μας να σχεδιάσουμε εκπαιδευτικά συστήματα που να είναι πολύτιμα, χρήσιμα για τα παιδιά, για τους νέους. Και να εξασφαλίσουμε στο μέτρο δυνατού ότι τα όσα συμβαίνουν στο πλαίσιο της ανώτητας εκπαίδευσης θα είναι επίσης πολύτιμα και χρήσιμα για τον κόσμο του σήμερα. Ένα ίδρυμα που ονομάζεται εκπαιδευτικό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι μέσα στο ίδρυμα αυτό προσφέρεται, παρέχεται γνώση. Αυτό πρέπει να το εξασφαλίσουμε. Και όχι μόνο για τον κόσμο της εργασίας, γενικά για την κοινωνία. Γιατί μέχρι τις τραγικές επιθέσεις του Παρισιού αναφερόμασταν στα έγγραφα της παιδείας στην απασχολησιμότητα χωρίς να αναφερόμαστε επίσης στην κοινωνία των πολιτών. Σήμερα καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να αναφερόμαστε στο σύνολο της εργασίας αλλά και της ζωής. Και αυτά τα δύο να μην είναι σε σύγκρουση μεταξύ τους. Κριτική σκέψη, δυνατότητα να, να κανείς ε, στα πολύ περίπλοκα ύδατα της ε, τεχνολογίας σήμερα και της αγορά τι εργασίες έτσι όπω έχει διαμορφωθεί. Θα δώσουμε λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία στο νέο θεματολόγιο των δεξιοτήτων. Θα δούμε και το πλαίσιο, το ευρωπαϊκό πλαίσιο των προσόντων για να κινηθούμε από κοινού όλα τα κράτη-μέλη μαζί σε αυτό το πεδίο. πλαίσιο το οποίο σήμερα πρέπει να επικαιροποιηθεί. Γιατί δεν πρέπει να μιλούμε μόνο για την ακαδημαϊκή οδό, για την μάθηση online και για άλλου είδους εμπειρία ε, κατάρτισης ή εκπαιδευτική που δεν αναγνωρίζεται ενδεχομένως από τα εκπαιδευτικά τα ακαδημαϊκά Ινστιτούτα. Και τα διάφορα κράτη-μέλη έχουν τα δικά τους συστήματα έχουν διαφορές μεταξύ τους. Πρέπει όλα αυτά να τα να προοδεύσουμε επ' αυτόν παραλλήλως. Έχουμε συζητήσει και για το Europass, ε, πρέπει να συζητήσουμε στους επόμενους μήνες για το πώς θα προχωρήσουμε και με αυτό το πολύ σημαντικό εργαλείο προκειμένου να καταχωρίζονται, να εγγράφονται επισήμως κάπως αυτά τα προσόντα, αυτό το πλαίσιο των δεξιοτήτων του κάθε δυντικού εργαζομένου. Αυτό θα πρέπει να το ενημερώσουμε γιατί έχει προχωρήσει ο κόσμος. Έχουμε σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις και το Europass μπορεί να βοηθήσει στη μετακίνηση των ανθρώπων μεταξύ θέσεων απασχόλησης. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την προσπάθεια των Σλοβάκων συναδέλφων πριν από μας. Και βεβαίως προσβλέπουμε πολύ και στη συνεργασία μαζί σας με τους συνομοθέτες προκειμένου όλα αυτά να υλοποιηθούν. Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο στο θεματολόγιο όπως το αναφέρουν και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου είναι η ιχνηλάτηση των νεαρών ανθρώπων που αποφυτούν. Γιατί αν έχουμε δεδομένα στοιχεία σχετικά με αυτούς μπορούμε αντιστοίχως να διαμορφώνουμε και τα εκπαιδευτικά μας συστήματα. Σχετικά με το πού έχουν βρει θέση απασχόλησης, αν έχουν βρει, πού έχουν τροφοδοτηθεί. Και βεβαίω θα εορτάσουμε και την 30η επέτειο του Εράσμου, γιατί αν έχουμε ένα πρόγραμμα που οπωσδήποτε έχει θετικά αποτελέσματα και θετικό αντίκτυπο συνολικά, θετική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει, είναι το Εράσμου. Θα πάω τώρα στις ε, πολιτικές για την νεολαία. Θα έχουμε πρωτοβουλίες με σαφείς στόχους μετρήσιμους στο βαθμό του δυνατού. Πρέπει να ενδυναμώσουμε την κατανόηση των νέων ε, για τη δημοκρατική κοινωνία των πολιτών, τη διαφορετικότητα και την πολιτιστική μεταξύ άλλων. Πρέπει να προετοιμάσουμε τους νέους μας να συμμετέχουν ενεργά σε ανοιχτές και δημοκρατικές κοινωνίες, ιδιαιτέρως τη στιγμή που αυτές οι αξίες πλήττονται αυτή τη στιγμή. Ήδη αναφέρθηκα στην διαμείου μάθηση και στην ανάπτυξη των προσόντων και των δεξιοτήτων είναι και αυτό σημαντικό. Δηλαδή όχι μόνο δεξιότητες επαγγελματικές αλλά δεξιότητες για την προσωπική ζωή του καθενός και για τη ζωή στην κοινωνία. Αυτά δηλαδή που θα επιτρέψουν στους νέους να είναι ενεργοί πολίτες και να έχουν και συνείδηση ως πολίτες. Επίσης οι εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας γνωρίζουμε και από την δική μας εσωτερική εμπειρία ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν τους νέους και στην προσωπική του ζωή και στην επαγγελματική του αδειοδρομία. Θα έχουμε λοιπόν, θα σχεδιάσουμε συμπεράσματα του Συμβουλίου σχεδιαστικά τη βοήθεια που μπορούμε να παράσουμε στους νέους για να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες ώστε να έχουν μια ομαλή μετάβαση από την σπουδαστική τους στην επαγγελματική του ζωή. Αυτά το Μάιο με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου δηλαδή. Και γνωρίζουμε πώς έχει τονιστεί το θέμα των ανακοινώσεων της ε, Επιτροπής ε, σχετικά με την νεολαία, ε, τα θέματα αλληλεγγύης που είναι επίσης πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες γιατί και αυτά βοηθούν τους νέους. Η συνολική θεματική προτεραιότητα για την περίοδο μέχρι τον Ιούνιο είναι το να επιτρέψουμε σε όλους τους νέους να συμμετάσχουν ενεργά σε μια διασυνδεδεμένη Ευρώπη και να είναι έτοιμοι για την κοινωνία. Θα έχουμε δύο σημαντικά συνέδρια στη Μάλτα, συναντήσεις, ένα διαφραμένο διάλογο 21 με 23 Μαρτίου, όπου περιμένουμε τους νέους εκεί για να εκφραστούν, να τοποθετηθούν μόνοι τους. Γιατί ένα από τα κοινά που έχουμε ως κράτος, τουλάχιστον, είναι όταν μιλούμε για τους νέους, όταν σχεδιάζουμε πολιτικές για τους νέους, συχνά το κάνουμε αυτό χωρίς να τους ακούμε, χωρίς να ακούμε τι έχουν να πούν εκείνοι. Είναι σημαντικό λοιπόν να τους ακούσουμε και ελπίζουμε ότι αυτό μπορεί να καταλήξει στον σχεδιασμό καλύτερων πολιτικών. Για τα θέματα αθλητισμού, τα οποία είναι πολύ σημαντικά πιστεύουμε, όχι μόνο για την σωματική αλλά και για την πνευματική υγεία. Θα προωθήσουμε τον εθελοντισμό μεταξύ άλλων στον αθλητισμό γιατί και αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και θα αναπτύξουμε μία από τις θεματικές που προκύπτει από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Ελπίζουμε ότι στο Συμβούλιο του Μαΐου θα συμπεριληφθούν και αυτά τα σημεία Προετοιμάζουμε και το πρόγραμμα εργασία για τα θέματα νεολαία και αθλητισμού επί τη βάση των ανακοινώσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και επίση, προσπαθούμε να αναπτύξουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τα, θέμα, για τα θέματα προσβασιμότητας, διακυβέρνησης και αθλητισμού. Η καταπολέμηση του ντοπαρίσματος. Έχουμε και τον Παγκόσμιο Οργανισμό της συνάντηση στο Μόντριελ. Θα, θα είμαστε εκεί για να παρουσιάσουμε τις απόψεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ζητήσω τώρα από τον συνάδελφο, από τον κύριο Μπονίτσι, να μας δώσει τα δικά του, τη δική του συνεισφορά για τα θέματα πολιτισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ Βαρτόλο. Θα ήθελα να δώσουμε το λόγο τώρα στον Υπουργό Μπονίτσι, που είναι Υπουργό Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λέει εδώ. Αλλά προφανώς ως Υπουργός Πολιτισμού παρευρίσκεστε και με χαρά θα ακούσουμε ε, τις προγραμματικές δηλώσεις και τα σχέδιά σας για το επόμενο εξάμεινο για τον πολιτισμό και τα μέσα ενημέρωσης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Κάμερβελτ. Θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ για την εκλογή σας στο νέο αυτό αξίωμα. Είστε πλέον πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, πολύ σημαντική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να συγχαρώ όμως και την κυρία Κώστα, για την θητεία της ε, μέχρι τώρα. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα αλλά και για τον συνάδελφό μου τον κύριο Μπαρτόλο να βρισκόμαστε εδώ πέρα. Πιστεύουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην εργασία την οποία καλούνται να διεξάγουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άποψή μας λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να διδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ίδια τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Και τι εννοώ όταν το λέω αυτό. Στην πράξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι σημαντική τόσο για τα σημαντικά ζητήματα, αλλά και για τα ζητήματα δευτερεύουσα σημασία. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι κάθε φορά που οι Ευρωπαίοι πολίτες ξυπνάνε το πρωί, πρωτού πάνε στη δουλειά ή αυτοί που πηγαίνουν στη δουλειά τους, οι άνθρωποι οι οποίοι ε, θέλουν να διασφαλίσουν καλύτερο επίπεδο εκπαίδευση για τα παιδιά του, οι άνθρωποι αυτοί που επιστρέφουν στο σπίτι του μετά από μια σκληρή μέρα εργασία και ξαναβρίσκουν την οικογένειά του, να είναι σε θέση πραγματικά να εκτιμήσουν σπουδαία ή λιγότερο σπουδαία πράγματα, τα οποία έχουν διασφαλίσει όμω για τη ζωή του τα ίδια τα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μπορούν να συνειδητοποιούν δηλαδή ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση βελτιώνει τελικά το επίπεδο διαβίωσή του. Αν υπάρχει λοιπόν ένας τομέας, ο οποίος πραγματικά επηρεάζει πολύ σημαντικά την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών, αυτός είναι σίγουρα ο τομέας του πολιτισμού. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για τόσα έκανε η Σλοβακική Προεδρία στον τομέα του πολιτισμού, κατά τη διάρκεια δηλαδή της δικής της Προεδρίας, και χαίρομαι πάρα πολύ βέβαια και για το θεματολόγιο και τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει εμείς ως Προεδρία, γιατί πιστεύω ότι οι στόχοι αυτοί πραγματικά θα επηρεάσουν άμεσα τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Θα ήθελα λοιπόν να σα παρουσιάσω εν συντομία τι προτεραιότητε τη Μαλτέζικη Προεδρία στον τομέα του πολιτισμού για του επόμενου έξι μήνε. Για άλλη μια φορά τονίζω ότι ο τομέα αυτό του πολιτισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή των ίδιων των Ευρωπαίων πολιτών. οι άνθρωποι οι οποίοι αυτοί παρακολουθούν τι κάνουμε στον τομέα αυτό. Ας ξεκινήσουμε με τον οπτικοακουστικό τομέα. Ξέρετε ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχαμε την εξή κατάσταση. Η τηλεόραση ρυθμίζεται από συγκεκριμένου κανόνες. Για παράδειγμα υπάρχουν κανόνες σύμφωνα με τους οποίους ένα συγκεκριμένο ποσοστό εκπομπών θα πρέπει να αφιερώνεται σε ευρωπαϊκές ταινίε. Έχουμε όμως και τα μέσα ενημέρωση στα επιγραμματικά, τα online, στο διαδίκτυο, τα οποία δεν ρυθμίζονται από συγκεκριμένους κανόνες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη πολυμορφία και πλουραλισμό ακόμα και στα επιγραμμικά αυτά μέσα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες μας πραγματικά προστατεύονται από οποιαδήποτε ρητορική μίσους, ότι προστατεύουμε επίσης τους ανήλικους από συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο θα μπορούσε να είναι βλαβερό για αυτούς και καταλαβαίνετε ότι η πτυχή αυτή θα είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι χρησιμοποιούν τα επιγραμμικά μέσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο 2016 υπέβαλε μια ανακοίνωση και στη συνέχεια το Συμβούλιο ξεκίνησε να επεξεργάζεται το πολύπλοκο αυτό κείμενο, προσπαθώντας επίσης να αποτιμήσει ποιες ήταν οι επιπτώσεις για τον ευρωπαϊκό οπτικακοστικό τομέα και τη σχετική αγορά. Τον Νοέμβριο του 2016 το Συμβούλιο Πολιτισμού και Νεολαίας ενέκρινε μία έκθεση που αποτιμεί την πρόοδο που έχει γίνει μέχρι στιγμής εντοπίζονται στα σημαντικότερα σημεία για το Συμβούλιο. Υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία είναι σημαντικά για το Συμβούλιο, εκ των οποίων το πιο σημαντικό θα έλεγα ότι είναι η επέκταση του πεδίου εφαρμογή και για τις πλατφόρμες ανταλλαγής βίντεο, όπως για παράδειγμα το YouTube, να θέσουμε συγκεκριμένου ορισμούς όσον αφορά την πλατφόρμα αυτή και να δούμε και σε ποιο επίπεδο θα μπορούμε να ρυθμίσουμε τελικά αυτή την πλατφόρμα ανταλλαγής ε, βίντεο. Ξέρετε ότι οι πλατφόρμες αυτές αυτή τη στιγμή δεν ρυθμίζονται από, τις οπτικοκουστικές, από την οδηγία οπτικοκουστικών υπηρεσιών. Θέλουμε επίσης να δημιουργήσουμε ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των παραδοσιακών μέσων και των νέων ψηφιακών μέσων. Και τρίτον, θέλουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία της χρησιμοποίησης, τη βελτίωση μάλλον της αρχής της χώρας προέλευσης. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η αρχή αυτή. Και τέλος, τίθενται και πάρα πολλά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τους μηχανισμούς παρακολούθησης και επίβλεψης, ζητήματα τα οποία πρέπει να αποσαφινιστούν. Για παράδειγμα, η παρατεταμένη χρήση της αυτορύθμισης ή να δούμε τι μπορεί να γίνει με τις εθνικές εθνιστικές ρυθμιστικές μπορεί να επισημοποιηθεί η ρυθμιστική ευρωπαϊκή ομάδα έργα όσον αφορά τι ευρωπαϊκέ ρυθμιστικέ αρχέ. Για όλα αυτά τα ζητήματα, σε συνεργασία με τι προηγούμενε Προεδρίε, προετοιμάσαμε μία σειρά από συμβαστικέ προτάσει, οι οποίε επί του παρόντο εξετάζονται από τι προπαρασκευαστικέ ομάδε εργασία του Συμβουλίου. Θα συνεχίσουμε την εργασία αυτή κατά τη διάρκεια τη δική μα Προεδρία και ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε μία συμφωνία στα πλαίσια του Συμβουλίου, ότι θα καταλήξουμε δηλαδή σε μια γενική προσέγγιση και ελπίζουμε ότι στα τέλη Μαΐου στο σχετικό συμβούλιο θα καταφέρουμε να εγκρίνουμε την προσέγγιση αυτή. Αν η προσπάθεια μας αυτή στεφθεί με επιτυχία, θα καταφέρουμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με εσά, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή, και αν είναι σωστέ οι πληροφορίε μου, πιστεύω ότι και εσεί ετοιμάζεστε και ότι θα είστε έτοιμοι την περίοδο αυτή. Προσβλέπω λοιπόν σε μια επικοδομητική συνεργασία μεταξύ ημών για το ζήτημα αυτό που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά μπορεί να επιφέρει πολλές βελτιώσεις στη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Έχοντας αυτά κατά νου θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο συγητές και την κυρία Κάμερβέτ και την κυρία Βερχόιν για την σημαντική εργασία που έχουν κάνει για την έκθεση αυτή όσον αφορά τις υπηρεσίες οπτικοκουστικών μέσων. Πρόταση που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και καθοριστική για τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχοντα μια επικοδομητική λοιπόν συνεργασία μεταξύ ημών, είμαι σίγουρο ότι θα καταφέρουμε να σημειώσουμε επαρκή πρόοδο για την πρόταση αυτή και θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή βάση, σε μια κοινή τοποθέτηση. Θα συνεργαστούμε επίση και με τι επερχόμενε προεδρίε προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε μια ομαλή διεξαγωγή τη πρόταση αυτή. Τώρα, στον τομέα του πολιτισμού υπάρχει μια πρόταση για, μια, για το Ευρωπαϊκό Έτο πολιτιστική κληρονομία 2018 και έχουμε επίση και το ζήτημα των ευρωπαϊκών πολιτιστικών πρωτευουσών όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που η Μάλτα έχει την ε, προεδρία του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της, ε, του εξαμήνου αυτού και θα είναι σε θέση κατά αυτόν τον τρόπο να προωθήσει την πρόταση αυτή που έχει υποστηρίξει τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο. γιατί είναι και σχετικό έτοιμο προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χαίρομαι που και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατάφεραν να εξασφαλίσουν μια διαπραγματευτική εντολή πάρα πολύ γρήγορα. Και κατά αυτόν τον τρόπο ήταν δυνατό να έχουμε τον πρώτο τριμερή διάλογο ήδη το 2016. Η ιδέα αυτή λοιπόν είναι καταπληκτική και όντως συμφωνώ ότι θα πρέπει το 2018 να αποτελέσει το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ήδη βρισκόμαστε σε στενή επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να προτιμάσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον επόμενο άτυπο τριμερή διάλογο για το σημαντικό αυτό ζήτημα. Προβλέπεται μάλιστα για τις 9 Φεβρουαρίου ο τριμερής αυτός διάλογος και προσβλέπουμε σε μια επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων μέσα σε εκπροσωπώντας το Συμβούλιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τζιάκονο και την κυρία Κώστα, τους δύο εισηγητές που έχουν κάνει μια πολύ σημαντική σκληρή εργασία για τον φάκελο αυτό. Πιστεύω ότι και εδώ θα πρέπει να συνεργαστούμε προκειμένου να υπερκεράσουμε οποιασδήποτε διαστάσεις απόψεων μπορεί να έχουν προκύψει και να καταφέρουμε να σημειώσουμε πρόοδο προκειμένου να καταλήξουμε τελικά σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία, προκειμένου στη συνέχεια υπηρεσίε Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι σε θέση να προετοιμάσουν το Ευρωπαϊκό Αυτό Έτο Πολιτιστική Κληρονομιά 2018. Πιστεύω πραγματικά ότι κατά τη διάρκεια του έτου αυτού θα καταφέρουμε να φέρουμε πιο κοντά του Ευρωπαίου πολίτε, να συνειδητοποιήσουμε ότι μοιραζόμαστε μια κοινή πολιτιστική κληρονομιά και θα καταφέρουμε κατά αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τι προκλήσει Τη πολιτιστική κληρονομιά για την Ευρώπη. Χαίρομαι πάρα πολύ όμω που μπορούμε να προωθήσουμε και μία ακόμα πρόταση, την πρόταση για, την Ευρωπαϊ... για τις ευρωπαϊκές πολιτιστικές ε, πρωτεύουσες. Η Βαλέτα θα είναι πολιτιστική πρωτεύουσα το 2018 και θα κάνουμε κάθε το δυνατό προκειμένου να καταφέρουμε να προωθήσουμε την πρωτοβουλία αυτή ορόσημο για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα του πολιτισμού. Ξέρω το 2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο από κοινού ενέκριναν μία απόφαση που επέκτηνε τις ευρωπαϊκές, το πλαίσιο μάλλον για τις ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες μέχρι το 2033. Ένα από τα νέα στοιχεία επιτρέπουν τώρα σε υποψήφιες χώρες ή δυνάμει υποψήφιες χώρες να συμμετέχουν στα προγράμματα δράσης κάθε τρία χρόνια. Πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να επεκταθεί η δράση αυτή ακόμα και στις χώρες ΕΖΕΣ και στην, στην Ορβηγία, την Ισλανδία και στο Λίχτενστάιν και θα συμφωνήσετε φαντάζομαι μαζί μου ότι οι χώρες αυτές αποτελούν εταίρους Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για πάρα πολλά χρόνια στο τομέα του πολιτισμού και ορισμένες ήδη συμμετέχουν στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Προκειμένου να καταφέρουμε λοιπόν να έχουμε μία τέτοια θετική συνεργασία και να επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο, το Συμβούλιο στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου ενέκρινε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επεκταθεί η γεωγραφική κάλυψη της δράσης, της δράσης αυτής στις χώρες ΕΖΕΣ και ΟΧ προκειμένου να καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερο την πρωτοβουλία για τις ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες και εκτός των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσβλέπω λοιπόν σε μια επικοδομητική συνεργασία με την Επιτροπή σας και για το ζήτημα αυτό και προσβλέπω μια θετική συνεργασία με την εισηγήτρια κυρία Ξέλα προκειμένου να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα επιτρέπει και στις χώρες σε ΟΧΚΕΖΕΣ να μπορούν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή. Στον τομέα του πολιτισμού επίσης θα επεξεργαστούμε και μια άλλη ωραία ιδέα που προτάθηκε σχετικά πρόσφατα, το να μπορούμε να χρησιμοποιούμε δηλαδή τον πολιτισμό σε ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο διπλωματίας. Θα ξέρετε ότι έχουμε και συμπεράσματα του Συμβουλίου όσον αφορά μια στρατηγική προσέγγιση για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις. Μακροσκελής ο τίτλος αυτός θα έλεγα και μια πολύ ωραία κατά τα άλλα πρωτοβουλία, σύμφωνα με την οποία οι Υπουργοί Πολιτισμού θα πρέπει να εγκρίνουν σχετική πρόταση κατά τη διάρκεια τη συνεδρίαση του Μαΐου. Εγώ προέρχομαι από τη Μάλτα, έχουμε μια συγκεκριμένη γεωγραφική θέση, καθώ επίση και μια γλωσσική πολιτισμική κληρονομιά που μα θέτει στην κατάλληλη θέση προώθηση τη ιδέα αυτή. Ότι ο πολιτισμό δηλαδή μπορεί να αποτελέσει γέφυρα για περαιτέρω διάλογο μεταξύ των κρατών σε διάφορες περιοχές. Επίσης θα βασιστούμε στην πολιτική συζήτηση που έλαβε χώρα το Συμβούλιο τον Νοέμβριο, όπου οι Υπουργοί καλωσόρισαν την προσέγγιση αυτή για μια πιο στρατηγική χρήση του πολιτισμού στις διεθνείς σχέσεις. Βάση της εργασίας μας βέβαια θα είναι η κοινή ανακοίνωση προς μια νέα στρατηγική για διεθνείς ε, πολιτιστικές ε, σχέσεις που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης τον Ιούνιο του 2016. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι και στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σημειώσετε και εσείς σημαντική επιτυχία στη συνεργασία που είχατε μεταξύ της δικής σας Επιτροπής και της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Ξέρω ότι από κοινού συνεργαστήκατε για το ζήτημα αυτό για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και προσβλέπω λοιπόν την υποβολή της κοινή σα θέση όσον αφορά τις διεθνείς αυτές πολιτιστικές σχέσεις και αν δεν κάνω λάθος είναι η κυρία Κώστα και ο κύριος Μπρόκ που θα επεξεργαστούν την κοινή αυτή έκθεση. Συμφωνώ επίσης με την έκθεση της κυρίας Ward που ανέκρινε τον Ιανουάριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά το διαπολιτισμικό διάλογο, τη διαπολιτισμική πολυμορφία και την χρησιμοποίηση της εκπαίδευσης για την προώθηση των κοινών πολιτισμικών αξιών. Αντιμετωπίζουμε στον παγκοσμιοποιημένο μας κόσμο κοινέ προκλήσεις. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλο και περισσότερο τον πολιτισμό ακόμα και σε εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεδομένου των νέων αυτών προκλήσεων λοιπόν που αντιμετωπίζουμε στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο μας κόσμο, ο ρόλος του πολιτισμού στις εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται όλο και πιο σημαντικός και για τον ίδιο τον τομέα του πολιτισμού αλλά και για τις προτεραιότητες στα πλαίσια των εξωτερικών σχέσεων μετά τις βαρβαρικές ε, επιθέσεις που είχαμε στην Συρία, στο Μάλι, στο Ιράκ, συντοποιούμε όλοι ότι η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν έχει να κάνει μόνο με την εξαφάνιση συγκεκριμένων μνημείων, έχει να κάνει με την εξαφάνιση της πολιτιστικής ταυτότητας, των αξιών, το οποίο κατ' επέκταση σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε ούτε να χτίσουμε το παρόν, ούτε να αρωματιστούμε το μέλλον. Αυτή τη στιγμή έχει εξαφανιστεί οποιαδήποτε πολιτιστική κληρονομιά ή οποιοδήποτε παρελθόν. Καλούμεθα λοιπόν να περάσουμε από μια θέση όπου απλώς χρησιμοποιούσαμε τον πολιτισμό προκειμένου να δείχνουμε προς τους ε, πολίτες τι κάνουμε στον τομέα αυτό. Σε μια κατάσταση λοιπόν πρέπει να επέλθουμε όπου θα συνεργαζόμαστε περισσότερο με τις υπόλοιπες χώρες προκειμένου να έχουμε πλέον κάποιες κοινέ δράσεις. Ας ξεχάσουμε λοιπόν αυτή την απαρχαιωμένη ιδέα στην Μάλτα χρησιμοποιούμε τη λέξη βιτρίνα. Ας μην χρησιμοποιούμε πλέον τον πολιτισμό απλώς για να προωθήσουμε κάποια ιστορικά μνημεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε από κοινού προκειμένου να έχουμε κάποιες ουσιαστικές δράσεις. Και αν το κάνουμε αυτό, πραγματικά θα αυξηθεί η πολιτιστική συνεργασία με διάφορες χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε το κατάλληλο πλαίσιο προκειμένου να κάνουμε τα επόμενα βήματα στο πλαίσιο των διεθνών αυτών πολιτιστικών σχέσεων του μέλλοντος. Το ζήτημα αυτό θα το συζητάσουμε και στα πλαίσια μιας συνδιάσκεψης πλαίσιο που θα λάβει η χώρα στη Μάλτα 8 και 9 Μαρτίου για τον τομέα του πολιτισμού και στη συνέχεια θα έχουμε και την συμμετοχή αξιωματούχων από την Υπουργεία Πολιτισμού και την Υπουργεία Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για τον συγκερασμό των δύο αυτών τομέων, πολιτισμός και εξωτερικές σχέσεις, εξωτερική πολιτική. Εγώ προφανώς ως υπουργό Πολιτισμού προσβλέπω σε μια θετική, ανοιχτή και αποτελεσματική συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και τους δύο υπουργού για την παρουσίαση αυτή που μας κάνετε. Τι δείχνει το πρόγραμμα της Μαλτέζικης Προεδρίας ότι είναι πάρα πολύ φιλόδοξο και σε πολλά σημεία συμπίπτει και με τις δικές μας προτεραιότητες εδώ της Επιτροπής. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο πρώτα στους συντονιστές και τις συντονίστριες των πολιτικών ομάδων για τρία λεπτά. Εκαστός παρακαλώ να τηρήσετε το τρίλεπτο. Μετά θα μιλήσουν και τα άλλα μέλη και θα απαντήσουν στο τέλος οι δύο υπουργοί. Η Σαπίνε Φερχάιεν έχει πρώτη το λόγο, συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους δύο υπουργούς ε, που βρήκαν το χρόνο να έρθουν στην Επιτροπή μας για να μας παρουσιάσουν τις προτεραιότητες και τα βασικά σημεία. Θα ήθελα να τονίσω και χαιρόμαστε ε, ως ε, και αυτά που λέτε για την νεολαία, ε, για ε, τα κηρύγματα μίσους, για τα οπτικοακουστικά μέσα, θα πρέπει να έχουμε ίδιες απαιτήσει και υψηλά πρότυπα προς όλους και για όλους. Αυτό ε, συνάδει με τις δικές μας απόψεις των δύο εισηγητριών. Θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα σε αυτό το θέμα, γιατί αρκετά περιμέναμε μέχρι να φέρει πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν χρειάζονται τώρα άσκοπες καθυστερήσεις και χρονοτριβές. Και πραγματικά θα χαρούμε αν μπορέσουμε να αρχίσουμε τον τριμερή διάλογο το Μάιο. Δεύτερον, Erasmus ε, Plus. Γίνονται πολλές συζητήσεις αυτό τον καιρό για επιπλέον δραστηριότητε που συζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σκέφτεται. Ε, εδώ δίνω αυτό το νέο σώμα εθελοντών. Εμείς διατρανώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι όλες οι νέες δραστηριότητες στο Erasmus Plus ε, δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον τρέχοντο προπολογισμό. Αν φτιάχνουν νέες δραστηριότητε που είναι πολύ ωραίες οι ιδέες και οι προθέσεις, ε, χρειάζονται ε, νέα χρήματα, γιατί έτσι κι είναι ε, υπερφορτωμένος ο προπολογισμό Έχουμε περισσότερα προγράμματα από τα χρήματα που ε, διαθέτουμε για να τα χρηματοδοτήσουμε. Λοιπόν, μην έχουμε κανένα κανιβαλισμό τώρα και αυτοματισμό να παίρνουμε από το ένα πρόγραμμα το δίνουμε στο άλλο. Ε, και παρακαλώ και προσβλέπω στην υποστήριξη του Συμβουλίου στην προσπάθειά μας αυτή. Άλλο θέμα. Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Θα παρακαλούσα επίσης γρήγορα να προχωρήσει ο τριμερής διάλογος, να συμφωνήσουμε κοινοβούλιο και συμβούλιο. Ήδη έχουμε καθυστερήσει και εκεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αδράνησε ε, μέχρι να δεήσει, να εγκρίνει αυτό το έτος, αλλά είναι πολύ γρήγορα το 2018 και δεν προλαβαίνουμε. Και θα πρέπει να δημιουργηθεί και μια βιώσιμη έτσι, ε, ε, πώς να το πω, δράση και ένα αποτέλεσμα ε, που να μην περιορίζεται το 2018 αλλά να διαρκεί και μετά το 2018. Άρα ε, όσο περισσότερο καθυστερούμε τόσο αργότερα ε, θα αρχίσουν να τρέχουν τα προγράμματα το 2018. Γιατί υπάρχουν και τα κράτη-μέλη και διοικήσεις που χρειάζονται λίγο χρόνο για να προετοιμάσουν και να υλοποιήσουν αυτά τα προγράμματα ιδέες μπορεί να υπάρχουν πολλές και καλές, αλλά ξέρω πάντα ότι ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός χωλαίνει όταν αρχίζεις ένα εξάμεινο πριν. Είναι σχεδόν ανεφάρμοστα τέτοια πράγματα. Όταν πρόκειται για ένα ετήσιο πρόγραμμα. Και θα πρέπει και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να κάνουν βήματα ε, ένας προς την κατεύθυνση του άλλου. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Η Σίλβια Κώστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους δύο υπουργού ε, για τα πολύ καλά τους λόγια και για την, ε, τις δύο τοποθετήσεις τους ε, που έχουν πολλά σημεία σύγκληση με τις δικές μας προτεραιότητες και με τη δική μας βούληση για τη διαμόρφωση των δικών μας θεματικών προτεραιοτήτων. Άκουσα και την τοποθέτηση του Προέδρου σας, του κ. Μουσκάτ, και νομίζω ότι νομίζω ότι θα μπορέσουμε και εμείς να στηρίξουμε και να έχουμε ένα πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας. Είπατε και εσείς ότι σήμερα η διάσταση του πολιτισμού ε, και της παιδείας θα πρέπει να ενισχυθεί και να είναι και μια απάντηση της Ευρώπης απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Είναι λοιπόν προφανές ότι και στο Συμβούλιο θα πρέπει να είναι πιο κεντρική σημασία σε αυτό το πεδίο από ό,τι υπήρξε μέχρι εδώ. Τώρα, εμεί ελπίζουμε το συντομότερο δυνατόν, όπω και εσεί αναφερθήκατε, Υπουργέ ε, Μπάρτολο, την ε, ανακοίνωση τη Ιεραρχικής Επιτροπής ε, για τον εξυγχρονισμό των δομών της ενότητας παιδείας και νομίζουμε ότι και στη δική σας Προεδρία αυτό θα καλυφθεί μαζί και με τα θέματα του θεματολογίου ε, για τα προσόντα. Εμείς έχουμε θυμίσει ότι το θεματολόγιο αυτό θα πρέπει να κινηθεί στο πλαίσιο της διαβίου μαθήσεως και να, έχει μια, να διατηρεί την επαφή δηλαδή με το πλαίσιο αυτό και όχι μόνο επαγγελματική κατάρτιση. Το Ευρωπάς επίσης μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και προσλέπουμε στη συζήτηση μαζί σας γιατί είναι σημαντικό. Ένα άλλο θέμα που ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι εμείς ζητήσαμε επαρλημένως από την Αρική Επιτροπή να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή ε, στο πλαίσιο του σχεδίου Juncker και για τις πλατφόρμες και για τα έργα και τη στρατηγική που αφορά στην παιδεία, στην ε, βιομηχανία του πολιτισμού. Νομίζω ότι εδώ έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η δράση που θα μπορούσατε να αναλάβετε. Η ψηφιακή κοινωνία των πολιτών και οπτικοακουστικές υπηρεσίες, όλα αυτά είναι συνδεδεμένα στρέφομαι εδώ περισσότερο στον ε, Υπουργό Μπονίτσι, ε, το ζήτημα με την ψηφιακή στρατηγική είναι καταρχάς προσοχή στο θέμα και το εκπαιδευτικό. Γιατί δεν είναι μόνο καταναλωτές, είναι πολίτες κυρίως αυτοί που λαμβάνουν τις υπηρεσίε αυτές. Και οι εισηγήτριές μας ασχολούνται με αυτό, αλλά το θέμα της προστασίας των αλήκων και της προστασίες των πραγματικών δικαιωμάτων και τη δημιουργικότητα συνολικά στα διαδικτυακά περιεχόμενα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και οι κοινωνικές πλατφόρμες θα πρέπει να λάβουν περισσότερη ευθύνη εδώ. Και ολοκληρώνω αμέσως. Εμείς ε, θα συζητήσουμε στην Επιτροπή ΑΦΕ, θα πρέπει να ε, δούμε λίγο τη διακυβέρνηση του όλου ζητήματο αυτού και βεβαίω το ευρωπαϊκό έτος τέλο. Το ευρωπαϊκό έτος ε, θέλουμε ε, να έρθουμε σε επαφή με το Συμβουλίο, να βρούμε ένα σημείο ισορροπίας. Ε, είναι οι πρώτε συναντήσει. ελπίζω όμως πάρα πολύ σύντομα να κλείσουμε. Καταρχά, οι πόροι λοιπόν, όπως και τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην επεξεργασία του έτους αυτού του Ευρωπαϊκού. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ, Χέλγα Τρουπέλ, από τους Πρασίνους. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Δύο σημεία. Πρώτον, Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με βλέπετε, εδώ κάθομαι. Μας είπατε ότι σας ενδιαφέρει πάρα πολύ η πρωτοβουλία αυτή, ότι ήδη την επεξεργάζεστε προκειμένου να θεσπιστεί όντω το αυτό και να ευοδοθεί. Ξέρετε όμως πως έχει και η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πρόβλημα με τον προπολογισμό. Αν πραγματικά θέλετε να καταλήξετε σε μια συμβαστική λύση, τότε το Συμβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να αυξήσει κάπως τον προπολογισμό προκειμένου πραγματικά το πρόγραμμα αυτό, η πρωτοβουλία αυτή όντω να ευοδοθεί. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίσω αν εσεί είστε σε θέση ω Προεδρία να ασκήσετε πίεση στο Συμβούλιο προκειμένου τελικά να καταλήξουμε όντω σε συμβαστική λύση Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, διεθνείς πολιτιστικέ σχέσεις. Το ζήτημα αυτό είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να δούμε λίγο και τη στρατηγική προσέγγιση δεν νομίζω ότι θα πρέπει απλώς να εξάγουμε τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, αλλά πώς μπορούμε πραγματικά να συνεργαστούμε στο πολιτιστικό τομέα με άλλες μη κυβερνητικέ οργανώσεις, με πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα. Επ' αυτού μπορείτε να κάνετε κι εσείς μια τέτοια προσέγγιση. Συμφωνείτε με την προσέγγιση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κανονικά τώρα ακολουθούν οι υπόλοιποι βουλευτέ, διαβάζω ονόματα. Μήπω ξέχασα κανένα. Λοιπόν, να κλείσω τον κατάλογο, μην ξεχάσω κανένα για να μπορέσουν να απαντήσουν και οι υπουργοί. Νέκαχ και Μπόσκορ, εννιά είμαστε. Ένα λεπτό πάει. Ένα λεπτό, τι να κάνουμε. Για να προλάβουμε και να απαντήσουν και οι υπουργοί μας. Η κυρία Κομοντίνη, παρακαλώ. Ναι, από το Ευρωπαϊκό Τσέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. η Υπουργή Μπάρτολο, ποια από τις θεματικές προτεραιότητες ε, προβλέπετε επί των θεμάτων παιδεία ότι μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο και πώς θα μπορέσει να συνεχίσει η δουλειά παρά τα σκάνδαλα διαφθοράς που έχουν πλήξει το Υπουργείο σας. Και αντί να δώσουμε άλλη μια συνέντευξη τύπου σχετικά με αυτά τα θέματα διαφθοράς, πώς θα μπορέσει να συνεχίσει λοιπόν η δουλειά ομαλά. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομη και συγκεκριμένη ερώτηση, κυρία Λεμπέτσκα. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα τα λόγια των Υπουργών και τους ευχαριστώ για τις εισηγήσεις τους. Συμφωνώ με τις προτεραιότητες που μας ε, περιέγραψαν. Έχω μια ερώτηση προς τον Υπουργό Μπάρτολο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να επιτύχετε αυτούς τους στόχους. Εκτός και αν συμπεριλάβουμε και τους διδασκάλους, τους καθηγητές. Και δεν άκουσα κάποια λόγια από εσάς, ε, σχετι... Ε, κάποια αναφορά στο πώς θα μπορέσουμε να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές, να περιλάβουμε τους διδάσκοντες σε όλο το πλαίσιο της διαδίου μαθήσεως. Ε, επίσης πρέπει να θυμίσω ότι τα πανεπιστήμια είναι αυτόνομοι φορείς, δεν μπορούμε να τους επιβάλλουμε κάποιο πρόγραμμα μαθήσεως. Εάν όμως ενός εργοδοτών θα μπορούσαν να υποβάλουν κάποιες προτάσεις, θα μπορούσαμε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον να τις υποβάλουμε, αν θέλετε, ως προτάσεις προς τα πανεπιστήμια. Πώς νομίζετε λοιπόν ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των πανεπιστημιακών φορέων. Ευχαριστώ πολύ κύριο Βέντα. Ευρωπαϊκό Ευχαριστώ πρόεδρε αξιότιμοι υπουργοί, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο για τις παρουσιάσεις που κάνατε εδώ. Η συνάδελφος πριν από λίγο αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Εράσμους. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά τα οποία είπατε εσείς. του προγράμματος Εράσμους. Ενδεχομένω να ακούσουμε λοιπόν από εσά λίγο περισσότερα πράγματα για τι προτεραιότητε του προγράμματο αυτού. Κινητικότητα των φοιτητών αποτελεί αυτό για εσά προτεραιότητα. Προτίθεστε να αναλάβετε ενεργό δράση προκειμένου να προωθήσετε πραγματικά την επέτειο αυτή του προγράμματο Εράσμου. Αναφερθήκατε επίση στον αθλητισμό. Ο τομέα αυτό με απασχολεί όλο ιδιαίτερο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε το τομεί όπω η προσβασιμότητα σε διάφορα αθλήματα και η καταπολέμηση του ντόπινγκ. Ξέρω ότι την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια θα ασχοληθούμε με την έκθεση Τάκουλα για την καλύτερη διαχείριση των αθλημάτων και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και τη συνιστόσα εκείνη που έχει να κάνει με τα στημένα παιχνίδια. Επομένως, η ερώτησή μου είναι η ακόλουθη. Τι βήματα προτίθεστε εσείς να ακολουθήσετε όσον αφορά την σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση των στημένων παιχνιδιών. Το ζήτημα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς που είμαστε ευρωβουλευτές. Θα θέλαμε πραγματικά κατά τη διάρκεια του 2017 να ασχοληθούμε εκ του σύνεγγυς με το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μίτση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. να ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία στους δύο αυτούς υπουργούς που έχουν πολύ σημαντικά χαρτοφυλάκια και τα οποία θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο επί των πολιτών και επί της ε, απασχόλησης και του πολιτισμού. Αυτή η Προεδρία δεν έρχεται σε μια εύκολη στιγμή, σε καμία περίπτωση. Ελπίζω όμως να αισθανθούν οι πολίτες μέχρι να ολοκληρωθεί το εξάμεινό της ότι θα έχουν κάτι ανακτήσει, κάτι κερδίσει. Σχετικά με τις ε, προτεραιότητες, αναφερθήκατε πάρα πολύ στο πλαίσιο των δεξιοτήτων, στο νέο θεματολόγιο, αλλά εδώ η Κομισιόν ε, δεν έχει δώσει πολύ μεγάλη σημασία θα έλεγα. Υπήρξε μια soft προσέγγιση αυτή. ένα σημαντικό ποσοστό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ε, θεωρούν ότι παρέχουν το κατάλληλο περιεχόμενο, ενώ ένα αντίστοιχο ποσοστό των εργοδοτών πιστεύουν πως όχι. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό, σε αυτή την εξισορρόπηση. Ε, επίσης η παιδεία είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και για να αναφερθώ και στο ερώτημα του συναδέλφου, σχετικά με το στήσιμο των παιχνιδιών, μήπως θα μπορούσε να μας εξηγήσει ο Υπουργός καθότι δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση ακόμα δεν είναι θέμα προτεραιότητας ε, το στήσιμο των παιχνιδιών για τη Μαλτέζικη Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργή, αναφερθήκατε σε διάφορες προτεραιότητες. Νομίζω ότι αν πραγματικά θέλουμε να σημειώσουμε επιτυχία θα πρέπει να περιοριστούμε σε συγκεκριμένες προτεραιότητες, οποίες ανέφεραν ορισμένοι συνάδελφοι. Επί της επεξεργασίας νομοθεσίας νομίζω ότι θα πρέπει να σημειώσουμε πρόοδο στην συζήτηση της για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειαζόμαστε επιγόντως μία νέα οδηγία η οποία θα ανταποκρίνεται στην εμφάνιση νέων τεχνολογιών και πολύ φοβάμαι ότι εδώ πέρα βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρκετά πίσω. Θα πρέπει επίση να καταφέρουμε να προστατεύσουμε τους νέους και τους ανήλικους από ακραίο περιεχόμενο ή περιεχόμενο μίσου, το οποίο βρίσκεται πολλές φορές στο διαδίκτυο. Θα πρέπει λοιπόν το πεδίο εφαρμογή να επεκταθεί και σε νέε ψηφιακέ πλατφόρμες. Θα πρέπει να τονίσουμε λοιπόν περισσότερο τα όσα θα γίνουν για τις υπηρεσίες οπτικοσκών μέσων και να ασχοληθούμε επίσης και με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υποβάλει την ιδέα αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να εμπλακούμε και εμείς προκειμένου να θεσπιστεί το έτος αυτό το συντομότερο δυνατό. Όσον αφορά το πρόγραμμα Εράσμους. Και πάλι εδώ πέρα θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα αυτό, προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει ομαλά. Και θα ασχοληθούμε και με το ζήτημα του στήσιματος των παιχνιδιών. Ευχαριστώ κύριε Μόργαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να προσθέσω και εγώ τις δικές μου ευχαριστίες στους υπουργούς μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Συμφωνώ και με τις προτεραιότητες και επ' αυτού θέλω απλώς να σχολιάσω για την απασχόληση και την παιδεία Επιτρέψτε μου να σας πω ότι με μεγάλη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή για την βιομηχανία του πολιτιστικού περιεχομένου αυτά ψηφίστηκαν το Δεκέμβριο τα λέω αυτά γιατί σε σχέση με την απασχόληση των νέων και για λόγους συντομίας είχαμε ε, ε, καθορίσει για πολλούς και διάφορους λόγους τέλος πάντων ότι ο τομέας αυτός δεν κάμφθηκε από την κρίση του 2008. Και εδώ πρέπει να επενδύσουμε χωρίς να περιμένουμε για να έχουμε αποτελέσματα. Και υπάρχει δέσμευση και του Πρόεδρου Γιούνκερ που μιλούσε για αναβιομηχανοποίηση της Ευρώπης από το 16% στο 20% του ΕΠ. Εδώ είναι ένας από τους τομείς που ζητήσαμε να είναι στρατηγική εστίαση για τις επενδύσεις. Επίσης εδώ έχουμε μια άμεση διασύνδεση με τον τουρισμό. 26 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης έχουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γουόρτ, πάλι σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για την αναφορά σας στην ε, γνωμοδότησή μου η οποία ανακρίθη πριν από ένα χρόνο στο Κοινοβούλιο και θα ήταν πάρα πολύ καλό να δούμε περισσότερες από τις συστάσεις αυτές να ενισχύονται και να ενσωματώνονται στις πολιτικές των κρατών μελών. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερα από εσά ιδιαίτερα για το ρόλο των καλλιτεχνών ως φορείς αλλαγής αντιλαμβάνεστε το σχετισμό μεταξύ των θεμάτων απασχόλησης και παιδείας, αλλά ο ρόλος των καλλιτεχνών είναι πολύ σημαντικός πιστεύω. Είναι άνθρωποι που μπορούν να ανανεώσουν την κοινωνία και την οικονομία μέσω της βιομηχανίας του πολιτισμού, αλλά είναι ακριβώς αυτοί οι φορείς της αλλαγής που επιθυμούμε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπόσκορ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για τις παρουσιάσεις. Πολύ χρήσιμα αυτά που ακούσαμε. Ο Υπουργό Μπάρτολο ε, μας μίλησε για τους δείχτες ε, της ενεργείας των νέων που παραμένουν πάρα πολύ χαμηλοί και ανεπαρκείς και τα προσόντα και οι δεξιότητες των νέων μας χωλένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ε, Προεδρία λοιπόν ε, έχει δηλώσει την πρόθεση να βελτιωθούν ε, αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Συγκεκριμένα ρωτώ και πώς θα το υλοποιήσετε αυτό. Υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες μέχρι το 2020. Εσείς πώς θα τη μεταφέρετε στην πράξη αυτή την πρόθεση. Και τι γίνεται με τις μειονότητες, αναφερθήκατε σε άτομα με αναπηρία ή τις σεξουαλικές μειονότητες, τι γίνεται με τις εθνοτικές μειονότητες και πώς θα τις ε, ε, προωθήσετε. Ευχαριστώ κύριος Νέκοφ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εξότιμοι Υπουργοί. Έχω να σας κάνω την εξής ερώτηση. Στο πρόγραμμα της Προεδρίας σας Είπατε ότι μία από τις προτεραιότητές σας είναι η απασχόληση των νέων. Η Μάλτα, τι είδους προσοχή έχει δώσει στην επίσημη και άτυπη εκπαίδευση, προκειμένου να καταφέρει να προωθήσει την εκπαίδευση στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, είπατε ότι θα δώσετε ιδιαίτερη σημασία στο νέο θεματολόγιο για τις νέες δεξιότητες. Τι συγκεκριμένα θα κάνετε όμως εσείς ως Προεδρία για το ζήτημα αυτό. Και τέλος, ευχηθώ κάθε επιτυχία στην Προεδρία σας. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια ε, και να υπογραμμίσω κάποια πράγματα. Και ως εισηγήτρια, η συνεισηγήτρια μαζί με τη Σαμπίνη Φερχάιεν, για την οδηγία για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες. Χαιρόμαστε και οι δύο πάρα πολύ που η Μαλτέζικη Προεδρία ε, από ό,τι φαίνεται έχει την πρόθεση να δώσει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή την ε, ε, έκθεση νομοθετικού περιεχομένου για να προχωρήσει στο Συμβούλιο και ελπίζω και στον τριμερή διάλογο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό και ελπίζουμε από όλες τις πλευρές ε, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο να έχουμε φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Ε, νομίζω ότι και οι δύο πλευρές καταβάλουν προσπάθειες και ελπίζω να τα καταφέρουμε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου σας. Για το Erasmus ε, Plus και το Σώμα Εθελοντών θα ήθελα να τονίσω ξεκάθαρα και ρητά ξανά κάτι που ακούσαμε προηγουμένως από τους συναδέλφους ότι έχουμε διατρανώσει ως Επιτροπή ε, ε, και συντεταγμένοι πάντα και ομόφωνα ότι όταν έχουμε νέες πρωτοβουλίες, νέα προγράμματα όπως είναι το Σώμα Εθελοντών που μπορεί να είναι ωραίο και καλό και χρήσιμο περιμένουμε συγκεκριμένες εξηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πώς θα χρηματοδοτούνται. Ή αυτό το Σώμα Εθελοντών πώς θα διαφοροποιείται ή πώς θα συνδέεται με ε, την Ευρωπαϊκή ε, Ειδική Υπηρεσία, θητεία ας πούμε, θελοντική θητεία. Και όταν φτιάχνουμε νέα προγράμματα θα πρέπει να βρίσκουμε και νέα χρήματα. Δεν φτάνουν τα λεφτά του Erasmus Plus για να χρηματοδοτούν όλες αυτές τις πρωτοβουλίες μας. Και παρακαλώ να τα διαβιβάσετε αυτά στο Συμβούλιο. Ε, αυτό είναι ακράδαντη πεποίθηση της πλειοψηφίας της Επιτροπής μας, ότι ε, νέες πρωτοβουλίες θα πρέπει να συνοδεύονται πάντα με νέα χρηματοδότηση και δεν μπορούμε να πετσοκόβουμε ε, άλλα προγράμματα που έτσι κι αλλιώς είναι σφιχτός ο προπολογισμό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το ίδιο ισχύει και για την πολιτιστική κληρονομιά. Θα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα, διότι ε, χρειάζονται ασφάλεια προγραμματισμού τα κράτη-μέλη. Το 2018 είναι πρώτον θυρών. Αύριο ξημερώνει 18. Τι θα γίνει, τα κράτη-μέλη δεν θα κανονίσουν τη πορεία τους, δεν θα προγραμματίσουν. Ακούω ότι είναι κάπως δύσκολη οι διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο και ελπίζω η Προεδρία της Μάλτας να βοηθήσει και ε, να απεμπλακεί κάπως η κατάσταση και να ε, δημιουργηθεί μια νέα δυναμική και από πλευράς ε, Συμβουλίου έτσι ώστε να έρθει σε αίσιο πέρας κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Ήθελα να σας τα πω και αυτά και τώρα σας παρακαλώ να απαντήσετε σύντομα στα σχόλια και τις παρατηρήσεις. Δεν ξέρω ποιος θέλει να αρχίσει, ο κύριος Μπάρτολο, ο κύριος Μπονίτσι, ε, όπως θέλετε. Παρακαλώ. Thank you. Thank you very much for... Ο κύριος Μπαρτόλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ενδιαφέρουσες αυτές ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Μα και πρωτού καν έρθουμε στη συνεδρίαση αυτή, γνωρίσαμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τη χρηματοδότηση του Erasmus Plus και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αλληλεγγύης και προφανώς για οποιαδήποτε νέα πρωτοβουλία θα πρέπει να υπάρχει και απαραίτητη χρηματοδότηση. Πάντως σας διαβεβαιώ ότι θα διαβιβάσουμε τις ανησυχίες αυτές και τις προτάσεις αυτές προς αρμοδίους. Ξέρουμε ότι ακόμα συζητείται βέβαια προπολογισμός για τα προγράμματα αυτά. Τώρα όσον αφορά τον εξυγχρονισμό της άτυπη εκπαίδευση Αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα και η κυρία Κώστα. Και έχουμε επίση και το θεματολόγιο των νέων δεξιοτήτων. Υπάρχει και το ζήτημα της διαβίου μάθηση. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι αλληλένδετα. Και αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον εγώ στο δικό μου το χαρτοφυλάκι ως υπουργό Παιδείας και Απασχόλησης συνειδητοποιώ όλο και περισσότερο ότι οι δύο αυτοί τομείς θα πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους. Το χείρημα δεν είναι εύκολο, πάντως ο μόνος τρόπος για να καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερο την ανώτατη εκπαίδευση και τη διαβίου είναι να καταφέρουμε να φέρουμε πιο κοντά τον τομέα της παιδείας και τον τομέα της απασχόλησης, έτσι ώστε να μπορούν οι νέοι οι οποίοι βγαίνουν από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης να βρίσκουν μια αξιοπρεπή εργασία στη συνέχεια. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό το πράγμα, τότε πολύ φοβάμαι ότι θα καταλήξουμε να έχουμε τελικά πανεπιστήμια τα οποία πολύ σύντομα θα είναι απλώς απαρχαιωμένα. Δεν γίνεται να λέμε ότι ε, έχουμε πανεπιστήμια 300, 400, 500 ετών και να ασχολούμεθα μόνο με την πολιστική αυτή κληρονομιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξακολουθούν τα πανεπιστήμια αυτά είναι σημαντικά και για το μέλλον. Περιμένουμε λοιπόν την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την υποβολή προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να καταφέρουμε να εξυγχρονίσουμε τους τομείς αυτούς. Και μέχρι την Άνοιξη πιστεύω ότι θα έχουμε καταφέρει να σημειώσουμε πρόοδο. Η χνηλασιμότητα στην οποία αναφέρθηκα είναι πάρα πολύ σημαντική. Μόνο αν καταφέρουμε να παρακολουθήσουμε την πορεία των πτυχιούχων, θα δούμε τελικά τι γίνεται στην πράξη στην αγορά εργασία. Ο καλύτερο μάλιστα τρόπο για να προσεγγίσουμε το ζήτημα αυτό είναι να έχουμε στενέ σχέσει μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κοινωνικών εταίρων και στη συνέχεια μεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε διάφορα επίπεδα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τα πάντα από τα πανεπιστήμια, γιατί πάρα πολλά πράγματα επιτελούνται και στον τομέα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όσον αφορά το Europass, θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε περισσότερο την πρόταση αυτή. Ακούστηκε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση όσον αφορά το ρόλο των διδασκόντων, των καθηγητών. Τα όσα συμβαίνουν στον τομέα της παιδείας δεν έχουν να κάνουν με τις δηλώσεις των Υπουργών Παιδείας, αλλά πολύ περισσότερο με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινή βάση στα πλαίσια των ε, τάξεων, των σχολείων και είναι πολύ σημαντικό να καταλήξουμε στην, στον απότερο αυτό στόχο που έχουμε θέσει, μια εκπαίδευση υψηλή ποιότητα για όλου. Αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από το ρόλο που δραματίζουν οι ίδιοι δάσκαλοι και οι καθηγητέ. Σε μια συνδιάσκεψη που έγινε πρόσφατα για το ζήτημα αυτό, καλέσαμε καθηγητέ και δασκάλου, οι οποίοι ήρθαν και μοιράστηκαν μαζί μα τη δική του την εμπειρία. Χρειαζόμαστε λοιπόν και εθνικά προγράμματα, καθότι το τομέα εξακολουθεί προφανώ και είναι ε, εθνική προτεραιότητα, ε, εθνική δικαιοδοσία, να έχουμε τη μεγαλύτερη συμμετοχή και των ίδιων των καθηγητών. Δεν θέλουμε μόνο συμμετοχή των καθηγητών από το πανεπιστημιακό επίπεδο, αλλά και στο επίπεδο τη δευτεροβάθμιας εκπαίδευση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τι συνθήκε προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν περισσότερο οι καθηγητές. Και νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε πολλά και από του ελβετού συναδέλφου πω κατάφεραν αυτοί να επικαιροποιήσουν το περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευση, στα πλαίσια τη ανώτερη εκπαίδευση, με αποτέλεσμα τελικά οι δεξιότητε των φοιτητών αντιστοιχούν όντω στις ανάγκες τη αγορά εργασία. Αυτό έγινε επειδή οι καθηγητέ πανεπιστημίου και εργοδότε, επιχειρηματίε ήρθαν από κοινού και κατάφεραν να συζητήσουν μεταξύ του για τι πραγματικέ ανάγκε στην αγορά εργασία. Και στη συνέχεια υπήρξε και ένα πρόγραμμα χρηματοδότηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών μονάδων, οι οποίε αντιστοιχούσαν πλέον στι πραγματικέ ανάγκε τη αγορά εργασία. Νομίζω ότι μπορούμε να διδαχθούμε πολλά από το πρόγραμμα αυτό, από αυτή την εμπειρία τη Ελβετία. Όσον αφορά το πρόγραμμα Εράσμου, προφανώ θέλουμε να εορτάσουμε την 30η επέτειο και αυτό μπορεί να γίνει μέσω των εκδηλώσεων που θα έχουμε στη Μάλτα και θα πρέπει να προσκαλέσουμε πιστεύω και όλους εκείνους ε, τους ε, φοιτητές που έχουν επιφεληθεί από το πρόγραμμα Εράσμου τα τελευταία 30 χρόνια οποίοι θα μπορούν να μας μιλήσουν οι ίδιοι για τη θετική εμπειρία που είχαν χάρη στο πρόγραμμα αυτό. Όσον αφορά τώρα ένα ευαίσθητο ζήτημα, το την καταπολέμηση του συστήματος των αθλητικών παιχνιδιών. Προφανώς θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τα φαινόμενα διαφθοράς στον αθλητισμό. Δυστυχώς όμως ε, τα στημένα παιχνίδια, το φαινόμενο αυτό σχετίζεται με την φορολογία την ίδια του τομέα του αθλητισμού και καταλαβαίνετε ότι ε, από μόνοι μας εμείς δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό. Όσον αφορά τώρα το θεματολόγιο, το θεματολόγιο δεξιοτήτων. Ο κύριος Μοργάνο αλλά και άλλοι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα και εμείς πιστεύουμε ότι ε, μόνο από κοινού μπορούμε να προωθήσουμε το νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη. Και το όλο αυτό ζήτημα συνδέεται και με το ερώτημα το οποίο θέσατε, τι θα κάνουμε εμεί ακριβώ στη Μάλτα κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα. Να καταφέρουμε δηλαδή να έχουμε πανεπιστήμια, τεχνικά πανεπιστήμια, τεχνικέ σχολέ, αλλά και σχολεία, δευτεροβάθμια δηλαδή εκπαίδευση, να συνεργαστούν μεταξύ τους προκειμένου να γνωρίζουν τελικά αν τα προγράμματα τα οποία παρέχουν, τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα όντως αντιστοιχούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σαφώς υπάρχουν αυτή τη στιγμή δεξιότητες και ικανότητες, υπάρχει ένα επίπεδο γνώσης, εμπειρίας, το οποίο λαμβάνεται εκτός τάξης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν οι έφηβοι να μπορούν να λαμβάνουν μια κάποια εμπειρία επαγγελματικής κατάρτισης μέσω προγραμμάτων άσκησης ή μαθητείας και εκτός σχολείου. Πρέπει αυτό να το έχουμε κατά νου. Και όσον αφορά πάλι το θεματολόγιο δεξιοτήτων, δεν διακυβεύεται μόνο εδώ πέρα το μέλλον εκατομμυρίων Ευρωπαίων, αλλά και το ίδιο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, αν δεν καταφέρουμε να πρικίσουμε με σημαντικές νέες δεξιότητες το εργατικό μας δυναμικό, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα είναι αγανακτισμένοι, Όλοι θα λένε ότι η παλαιά οικονομία πέθανε, αλλά ότι η νέα οικονομία θα τους προσφέρει νέες ευκαιρίες και καταλαβαίνετε πόσες δεινές επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των διαφορετικών τομέων να καταφέρει να συντονίσει τις πολιτικές της. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε μία ενιαία φωνή. Δεν γίνεται να λέμε διαφορετικά πράγματα όσον αφορά τον πολιτισμό και την παιδεία και να μιλάμε έπειτα εντελώς διαφορετικά, ή να έχουμε διαφορετική προσέγγιση όταν μιλάμε για χρηματοδότηση, για δημοσιονομική πολιτική σε καμία περίπτωση θα πρέπει οι αποφάσεις που λαμβάνουμε στο επίπεδο του προπολογισμού να βαίνουν κατά της ίδιας της κοινωνικής μας πολιτικής. Κοινωνική και οικονομική πολιτική θα πρέπει να βαδίζουν από κοινού. Οι δύο αυτοί τομείς, όπως γνωρίζετε, αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοεξαρτώνται και πραγματικά διακυβεύεται το ίδιο το ευρωπαϊκό μοντέλο. Τέλος. Ένα από τα επιγρεύματά μας μέχρι τον Ιούνιο ελπίζω ότι θα είναι οι συστάσεις του Συμβουλίου όσον αφορά την εκπαίδευση υψηλή ποιότητος για όλους. Θα έχουμε συμπεράσματα δηλαδή του Συμβουλίου όσον αφορά την πολυμορφία, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη. 25 χρόνια είμαι βουλευτή στη Μάλτα και ανέκαθεν έδιναν αγώνα κατά της διαφθοράς και αυτό προτίθεται να κάνουμε και στο μέλλον και δεν διστάζω να πάρω αποφάσεις σημαντικές κάθε φορά που βλέπω ότι ακόμα και στενοί συνεργάτες μου μπορεί να μην ακολουθούν, να θέλετε, το σωστό δρόμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε συγκεκριμένα υψηλά πρότυπα στα πλαίσια της πολιτικής ζωής, ιδίως όσον αφορά, για παράδειγμα, τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, αλλά δείτε λίγο την πορεία μου μέχρι σήμερα και θα λάβετε μια απάντηση στο ερώτημά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μπονίτσι τώρα. Έχετε το λόγο για να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις που σας έγιναν. Ελπίζω να έχω περισσότερο από ένα λεπτό, Πρόεδρε. Δύο λεπτά. Μου κάνει εντύπωση πώς μπορείτε εσείς να χειρίζεστε τα μόνο λεπτά. Τέλος πάντων. Να μην μακρηγορήσω, να μην καθυστερώ. Έχετε περισσότερο χρόνο, λέει η Πρόεδρο εκτό μικροφώνου. Ωραία, χαίρομαι Πρόεδρε. Με ικανοποιεί πολύ η συζήτηση που έγινε σήμερα και αν ήταν να γράψω μία αναφορά, μία έκθεση για τη σημερινή συζήτηση, θα έλεγα λιγότερα λόγια, περισσότερη πράξη. Γιατί κατάλαβα το μήνυμα που το Κοινοβούλιο διαβιβάζει και στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα για δύο χαρτοφυλάκια πολύ σημαντικά που έχουμε, που, θα, που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των πολιτών προς το καλύτερο. Την οδηγία υπηρεσιών για τα οπτικοακουστικά με μέσα και για την πολιτιστική κληρονομιά. Για τα οπτικοακουστικά μέσα και την οδηγία υπηρεσιών ακούσαμε τα σχόλιά σας τις παρατηρήσεις σας. Εγώ έχω μία μικρή κόρη, 8 χρονών, της αγόρασα μία τηλεόραση τον περασμένο Σεπτέμβριο, μία καινούργια τηλεόραση και της είπα ορίστε το χριστουγεννιάτικο δώρο σου. Μου, μου είπε δεν τη χρειάζομαι αυτή, έχω το iPad, έχω το, τον υπολογιστή μου, τι το χρειάζομαι. Αυτή είναι η πραγματικότητα που έχουμε σήμερα για μια οκτάχρονη ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι ασφαλής όταν ψάχνει το ίντερνετ, όταν κοιτάζει διάφορες ιστοσελίδες. Εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω και ως πατέρας αλλά και ως πολιτικός. Αυτό χρειαζόμαστε με την οδηγία των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όταν τα παιδιά μας είναι στο διαδίκτυο και κοιτάζουν διάφορες ιστοσελίδες θα υπάρχουν μηχανισμοί που θα προφυλάσσουν, θα φιλτράρουν το περιεχόμενο και θα προφυλάσσουν τα παιδιά μας. Εξού και η ευθύνη των παρόχων. Η οδηγία όμως είναι πολύ περισσότερο από αυτό. Αφορά και τα μηνύματα μίσους. Είμαι και υπουργό αρμόδιος για θέματα δικαιοσύνης. Θα είμαι και στο Συμβούλιο Τζάι και όταν συζητήσουμε με τους ε, συναδέλφους θα συζητήσουμε το θέμα αυτό των μηνυμάτων μίσους και θα του δώσουμε μεγάλη σημασία γιατί αυτό έχει άμεση σχέση με την ε, ριζοσπαστικοποίηση που είναι πολύ συχνά αποτέλεσμα της χρήσης, της κατανάλωσης κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Πρέπει να προστατεύσουμε τις κοινωνίες μας, αλλά πρέπει να καλύψουμε και ένα κενό ασφάλειας που υπάρχει. Η δέσμευσή μας λοιπόν ως Προεδρία της Μάλτας είναι ότι θα προχωρήσουμε το φάκελο αυτό όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Και για την οδηγία υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων σήμερα έχουμε μια κατάσταση και την οποία μια σειρά από ευρωπαϊκές παραγωγές μπορεί να προωθούνται στην τηλεόραση ενώ στο Netflix που η νεολαία χρησιμοποιεί καθημερινά δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εάν θέλουμε να προστατεύσουμε λοιπόν να καλλιεργήσουμε τη δημιουργική οικονομία όπως είπαν και οι συνάδελφοι γιατί να έχουμε ένα κανόνα στην τηλεόραση για ένα ελάχιστο ποσοστό ευρωπαϊκής παραγωγής που εμείς θεωρούμε ότι είναι καλός κανόνας, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε παραγωγούς όπως το Netflix. Χρειάζεται λοιπόν να εξισορροπήσουμε και αυτά, και αυτές τις αποκλήσεις. Πρέπει να κινηθούμε ταχαίως στο πλαίσιο της οδηγίας, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι και στο Netflix μεταξύ άλλων θα υπάρχει μία ποσόστοση περιεχομένου που θα προέρχεται από τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο, για παράδειγμα. Το οποίο θα είναι σημαντικό για τους καλλιτέχνες μας. Υπάρχει μια ρομαντική έτσι, ερμηνεία της τέχνης και των καλλιτεχνών. Εγώ λατρεύω το πεδίο της τέχνης, αλλά είναι και μια οικονομική πραγματικότητα ο τομέας της τέχνης και δημιουργεί και αυτός θέσεις απασχόλησης. Και αυτό καμιά φορά το ξεχνούμε. Μιλούμε και για την απασχόληση και σε αυτόν τον ανταγωνιστικό κόσμο πρέπει οι καλλιτέχνες και οι άνθρωποι που ζουν από τον τομέα της τέχνης να έχουν και αυτοί αντίστοιχες ευκαιρίες και στο διαδίκτυο και στα online περιεχόμενα. Πρέπει λοιπόν να κινηθούμε ώστε να διασφαλίσουμε τις διατάξεις της οδηγίας αυτής και σε αυτό το επίπεδο. Για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς που αρκετοί αναφερθήκατε, πρέπει να ομολογήσω ότι εδώ έχω μια κάποια σύγκρουση συμφερόντων, γιατί η Βαλέτα θα είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα το 18 και επομένως από όλους τους ανθρώπους στην αίθουσα εγώ είμαι εκείνος που θα ήθελε το 18 να είναι και έτος πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη την Ευρώπη που θα ήταν λιγότερο κύριος για τη βαλέτα αν θέλετε να το δει κανείς έτσι. Εν πάση περιπτώσει εμείς είμαστε απολύτως δεσμευμένοι πέρα από τα αστεία να προχωρήσουμε στο φάκελο αυτό και αντιλαμβανόμαστε βεβαίως και τις ανησυχίες που έχει υποβάλει το Κοινοβούλιο και εξερευνούμε διόδους, δυνατότητες ώστε να κινηθεί προς τα εμπρός το έργο αυτό. Και ότι το έργο αυτό θα έχει και κατάλληλη επαρκή χρηματοδότηση μαθαίνω ότι το Συμβούλιο επί της αρχής συμφωνεί με το Κοινοβούλιο ότι μπορεί να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση από υφιστάμενα μέσα κονδύλια. Αλλά περιμένω να ακούσω τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επ' αυτού. Σας βεβαιώνω λοιπόν ότι παρακολουθούμε το θέμα με μεγάλο ενδιαφέρον. πολλά θέματα ελέγχθησαν και σας ευχαριστώ για τις συνεισφορές σας. Τα τελευταία μου λόγια για... είναι αφιερωμένα σε αυτήν την ε, πολιτιστική διπλωματία. Συμφωνώ με τη Σίλβια που λέει ότι αν κάνουμε μια προσπάθεια, την κάνουμε από κενού με άλλες χώρες ώστε να εξασφαλίζουμε ότι θα έχουμε επαρκείς δομές διακυβέρνησης. Ότι θα έχουμε δώσει δηλαδή όλες τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες ώστε η προσπάθειά μας να καρποφορήσει. Θα το διαβάσω λοιπόν αυτό το σημαντικό μήνυμα στους συναδέλφους ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα καλλιεργήσουμε αυτό το πολύτιμο εργαλείο της πολιτιστικής διπλωματίας και θα εξασφαλίσουμε και τις επαρκείς δομές διακυβέρνηση. ώστε να είναι βέβαιο ότι κάθε ευρώ που προέρχεται από τους φορολογμένους να χρησιμοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να χάνουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την ε, πολύ καλή συζήτηση που είχαμε εδώ με τους εκπροσώπους της ε, Προεδρίας Μάλτας, με τους δύο υπουργού. Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μας αφιερώσατε εδώ σήμερα για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων για να είμαστε έτοιμοι. Πρόκειται για έργα και πρωτοβουλίες πάρα πολύ φιλόδοξα ώστε εντός του εξαμήνου να υλοποιηθούν, να στεφθούν με επιτυχία. Εξ όλων των μελών της Επιτροπής μας σας βεβαιώνω ότι μπορείτε να βασιστείτε στη δική μας υποστήριξη και συνεργασία και θα έλεγα ενεργό αλληλεγγύη από πλευράς μας, έτσι θα την έλεγα. Είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε και είμαι βέβαιη ότι θα ξανασυναντηθούμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία για το υπόλοιπο του εξαμήνου.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχουμε ακόμα τελειώσει, έχουμε ακόμα σημεία στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε ακόμα δύο σημεία για το πρωινό. Θα μπορούσα να σας ζητήσω παρακαλώ εκείνοι που θέλουν να εγκαταλείψουν την αίθουσα να το κάνουν ταχαίως και ησύχω ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμός. Πάμε λοιπόν στα δύο τελευταία σημεία της ημερησίας διατάξεως. Πρόκειται για την ε, εφαρμογή της συμφωνίας του Μαρακές. Όχι, όχι. Μάλλον διακόπτει η πρόεδρος και λέει σας παρακαλώ στα αγγλικά αν θέλετε να εγκαταλείψετε την αίθουσα γιατί πρέπει να συνεχίσουμε εμείς τη δουλειά εδώ. Το 17 λοιπόν σημείο είναι οι επιτρεπόμενες χρήσεις ε, ή άλλων αντικειμένων προστατεύονται από δικαιώματα δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα προ όφελο των τυφλών αμβλιόπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωση εντύπων. Κεντροποίηση οδηγία 2001-29 για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματο δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία τη πληροφορία. Η κυρία Τρούπελ θα μας κάνει με βέβαια μια εισαγωγή τώρα για να μας εξηγήσει ποιος είναι ο στόχος του φακέλου. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάντε μόνο λίγο ησυχία σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, να κάνω μια σύντομη εισαγωγή. Έχουμε τη συνθήκη του Μαρακές που εγκρίθηκε το 2013 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 60 περίπου χώρες έχουν υπογράψει τώρα τη σύμβαση αυτή, συμπεριλαμβανομένης τη ευρωπαϊκή Ένωσης. Είναι λοιπόν σαφές για μένα ότι υπάρχει μια δέσμευση προκειμένου να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα αυτό το οποίο έχει προκύψει. Τι μα ζητά λοιπόν η συνθήκη του Μαρακές. Λέει ότι τα συμβαλώμενα μέρη θα πρέπει να έχουν ε, υποχρεωτικέ εξαιρέσει και περιορισμού όσον αφορά τα δικαιώματα δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα ιδίω όσον αφορά προ όφελο των ε, τυφλών και των ατόμων που έχουν προβλήματα όρεση, προκειμένου να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να χρησιμοποιούν βιβλία σε άλλου εναλλακτικού μορφότυπου, για παράδειγμα μέσω τη γλώσσα Braille ή μέσω εχογραφημένων βιβλίων, audiobooks κτλ. Ουσιαστικά, κατά αυτόν τον τρόπο, θα σταματήσει η έλλειψη αυτή βιβλίων που έχει εντοπιστεί για τους τυφλούς και τα άτομα με προβλήματα όρασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο 5% των δημοσιευμένων βιβλίων είναι διαθέσιμα για άτομα με προβλήματα όρασης. Και αυτό αποδεικνύει ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει μια πραγματική αγορά για παρόμοια τέτοια έργα. Η συνθήκη του Μαρακές λοιπόν αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της πρόσβασης αυτών των ατόμων σε πολιτιστικές και εκπαιδευτικές πληροφορίες όπως κάθε άλλος πολίτης. Ξέρετε ότι οι υπόλοιποι πολίτες μπορούν να πάνε σε οποιαδήποτε βιβλιοθήκη και να βρουν εκεί πέρα έντυπα και βιβλία. Για έναν τυφλό όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, γιατί ακόμα και στις εξειδικευμένε αυτέ βιβλιοθήκε για του τυφλού δεν υπάρχουν τα απαραίτητα έργα ή απαραίτητο αριθμό έργων. Γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε μέσω τη πρώτη αυτή οδηγία να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη αυτή έργων και βιβλίων, προκειμένου τυφλοί ή αμβλίωπε να μπορούν τελικά να έχουν πρόσβαση στην ίδια πολιτιστική πολυμορφία και στον ίδιο πολιτιστικό πλούτο. Ξέρετε επίση ότι ε, οι προβλεπόμενες εξαιρέσεις, οι περιορισμοί ισχύουν μόνο για ένα πολύ περιορισμένο κύκλο προσώπων και μόνο για μη εμπορικού σκοπού. Υπάρχουν συγκεκριμένε προποθέσει, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες έργων. Και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις ελλείψεις που είδαμε αυτή τη στιγμή στην αγορά και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε βέβαια να περιορίσουμε την σχετική αγορά βιβλίων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ισχύουν συγκεκριμένοι μορφότυποι όπως η γραφή Braille ή Daisy και επομένω τα βιβλία αυτά δεν θα ανταγωνίζονται με τα έργα που προορίζονται για άτομα με κανονική όραση. Μιλάμε για διαφορετικά προϊόντα. Κατά την άποψή μου λοιπόν δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι οι εξοδοτημένε οντότητε που παράγουν αυτές τις προσβάσιμες μορφές εντύπων μπορούν τελικά να βλάψουν τους κατόχους δικαιωμάτων ή τους εκδότες μέσω της πειρατείας. Και επίσης η συνθήκη δεν πρόκειται να υπονομεύσει τη συνθήκη της συνήθεις να υπονομευσει τη συνθηκη της συνηθεις και δεν θα εμποδίσει τους κατόχους δικαιωμάτων από την αύξηση του αριθμού των τίτλων που παρέχονται σε κανονική μορφή. Δεν προωθεί τον εμπορικό ανταγωνισμό στον, εκδοτικό κλάδο και πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η συνθήκη υπάρχει λόγω του ότι η αγορά αυτή απέτυχε να καλύψει τα τυφλά ή με μειωμένη όραση άτομα. Ω εκ τούτου όλα τα αναγκαία μέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία και κατάλληλη εφαρμογή τη συνθήκη και καλό λοιπόν την ταχεία κύρωση τη συνθήκη του Μαρακέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να τονίσω για μία ακόμη φορά ότι ε, σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιο κίνδυνο όσον αφορά τα δικαιώματα του δημιουργού ή το δικαίωμα του copyright. Προφανώ προστατεύω αυτά τα δικαιώματα και θέλω να προασπιστούν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ορισμό όσον, όσον αφορά του τις εξοδοτημένες οντότητες, μόνο αυτές μπορούν να διαβιβάσουν για μη εμπορική χρήση τους νέους αυτούς μορφότυπους των βιβλίων. Τονίζω, δεν πρόκειται για νέα εμπορική χρήση των βιβλίων αυτών, πρόκειται για νέους μορφότυπους εναλλακτικού που παρέχονται για τυφλά άτομα ή τα άτομα που έχουν ειδικέ ανάγκες, προορισμένη όραση κτλ. Στόχος μας λοιπόν θα πρέπει να είναι να μην δημιουργήσουμε ένα νέο γραφειοκρατικό άχθος όσον αφορά τις κοινότητες αυτές των τυφλών που ήδη αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα. Ένα 5% μόνο των δημοσιευμένων βιβλίων είναι διαθέσιμα σε εναλλακτικέ μορφές, σε εναλλακτικού μορφότυπους. Θα ήθελα λοιπόν να καταφέρουμε να ακολουθήσουμε τους στόχους της προτινόμενης αυτής οδηγίας. Όσον αφορά τη διαδικασία αυτή καθεαυτή, το θίξαμε και το ζήτημα αυτό χθε. Πέτρε, θα μιλήσει με του αρμόδιου συναδέλφου. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε πολύ γρήγορα να καταλήξουμε σε μια καλή λύση, γιατί η φυστάμενη κατάσταση που ισχύει για του τυφλού ή για τα άτομα που έχουν περιορισμένη όραση είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι πραγματικά αφόρητη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να το πω εξ ονόματο όλων. Όλοι ενδιαφερόμαστε να προχωρήσουμε γρήγορα και να έχουμε και αποτελέσματα αρκετά σύντομα. Ε, όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Λοιπόν, τώρα έχω τη Σαμπίνη Φερχάιεν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να εκπροσωπήσω το δικό μας σκιώδη εισηγητή που δυστυχώς κολλείται και μου έχει δώσει μια δήλωση που θα διαβάσω εξ ονόματός του και για την έκθεση αυτή και την επόμενη. Χαίρομαι που επιτέλου συζητούμε στο Κοινοβούλιο την ε, οδηγία και τον κανονισμό για τη συνθήκη του Μαρακές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για ανθρώπου με ε, προβλήματα στην όραση που δεν μπορούν να διαβάσουν ε, έντυπα. Ε, υπάρχουν πολλοί φραγμοί και πολλά εμπόδια για τους ανθρώπους αυτούς, βιβλία γιατί προστατεύονται από copyright. Ε, αυτό που συζητούμε σήμερα στοχεύει στο να υπεραστούν αυτά τα εμπόδια, να υπάρξει ε, αλλαγή βεβαίως χωρίς να ζημιώνονται οι εκδότες ή ε, συγγραφείς και κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων. Η γρήγορη έγκριση του οδηγία και του κανονισμού Σαμπίνε σε διακόπτω. Μου ανάβει ένα λαμπάκι εδώ γιατί δεν σε προλαβαίνουν οι διερμηνείς. Ναι, διαβάζω γρήγορα. Ναι, ζητώ συγγνώμη από τις μεταφράστριες. Η γρήγορη λοιπόν έγκριση είναι απαραίτητη έτσι ώστε να τεθεί σε ισχύ η συνθήκη του Μαρακές. Γενικώ συμφωνώ ε, με τη θέση της εισηγήτριας και το γεγονός ότι θα πρέπει και τα δύο έγγραφα να ευθυγραμμιστούν με τη συνθήκη του ε, Μαρακές ε, για τους δικαιούχους ε, και την ε, δικαιούχο αρχή. Τα έγγραφα αυτά ε, είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους και γι' αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους ίδιους ορισμούς και την ίδια ορολογία. Αυτά ευχαριστώ πολύ. Η Ευχαριστώ πολύ, Χέλγα, για τη δουλειά που έχει κάνει για αυτό το θέμα. Ε, και πραγματικά χρειάζεται να εφηγραμμιστούν η οδηγία και ε, ο κανονισμός. Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην πλήρη ε, συμμετοχή στην ζωή και στην πνευματική ζωή και στην πολιτιστική. Αυτό είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Ήταν ορόσημο η συνθήκη του Μαρακές και περιμένουμε νέες κινήσεις. Εγώ μίλησα με πολλούς ε, εκπροσώπους ατόμων με αναπηρία, με πολλούς εκδότες, με πολλούς ε, εκπροσώπους ε, συγγραφέων και θα πρέπει να είναι σωστή η διατύπωση των κειμένων που εγκρίνουμε έτσι ώστε να εφαρμόζεται σωστά και η συνθήκη του Μαρακές εν ώψη της κύρωσης. Δηλαδή, άλλο είναι απειρία, άλλο είναι μια δυσκολία που έχει κάποιος πρόσβαση, γιατί είναι συγκεκριμένη η ε, αναφορά που γίνεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ότι ανάπηρο σε κάνει κοινωνία. Δεν είναι επειδή έχει ένα πρόβλημα σε ανάπηρο από μόνο σου. Είναι ένα θέμα διάδραση και αντίδραση των άλλων ε, σε μια δυσκολία, ένα πρόβλημα που έχει εσύ. Ε, ε, δηλαδή θα πρέπει να προσέξουμε την ορολογία μας Θα πρέπει να είμαστε πιο ειδικοί, πιο συγκεκριμένοι και να φέρουμε ότι, ε, ότι η συγκεκριμένη αρχή έχει να κάνει και με την πιστοποίηση και με την πίστη. Δηλαδή θα πρέπει τα ε, έργα που δημοσιεύονται να έχουν μια σταθερή ποιότητα και μια, ε, έναν έλεγχο. Η κοινωνία των πολιτών λοιπόν τι λέει για όλα αυτά. Συνάντησα κάποιον σε ένα φόρουμ ε, αναπηρίας και μου ανέφερε την προσωπική του εμπειρία. Ε, είναι τυφλός ο άνθρωπος, έχει ένα πρόβλημα όρασης και πραγματικά κατάλαβα από όλα αυτά που μου είπε το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χιμένες Μπαρμπάτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία σε αυτόν τον πολύ σημαντικό φάκελο. Να θυμίσω ότι η χώρα μου ήταν μία από τις πρώτες που επικύρωσε τη συμφωνία του Μακρακές ε, τον Μάιο του 2016. Οι τροπολογίες ε, που προτείνει η συγγήτρια για την οδηγία και για τον κανονισμό συμπεριλαμβανομένων και άλλων αναπηριών, εκτό των οπτικών δηλαδή, είναι πολύ σημαντικέ, Με ανησυχούν όμως κάποιες τροποποιήσεις ε, σχετικά με τις ε, εξουσιοδοτημένες αρχές που είναι ε, φορείς και οργανισμοί που έχουν ορίσει οι κυβερνήσεις αλλά και σε άλλο επίπεδο οργανισμοί μη κυβερνητικοί και στην οδηγική και στον ε, ε, κανονισμό αναφέρονται, ε, αναφέρονται οι διατάξεις σε φορείς μη κερδοσκοπικούς και άλλους. Η συνθήκη, η σύμβαση εστιάζεται όχι μόνο στα πνευματικά δικαιώματα, στα δικαιώματα δημιουργού, αλλά και δικαιώματα στη χρήση, στην ανάγνωση που έχουν σχέση με θεμελιώδη δικαιώματα και μεταξύ των οποίων και το δικαίωμα στην παιδεία. Τα ε, βιβλία σε ε, ακουστικό περιεχόμενο για παιδιά δηλαδή που έχουν προβλήματα οπτικά 30 εκατομμύρια ε, πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με προβλήματα στην όραση περιμένουν τις διατάξεις αυτών των νομοθετημάτων και είναι σημαντικό κυρία Σόιντροβα και μετά να περάσουμε στην έκθεση Τζαμπάτσκι και να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους δύο εισηγητές μαζί. Γιατί είναι λένετε αυτά τα δύο θέματα. Η κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Υποστηρίζω και εγώ την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την έκθεση φυσικά, ε, όπως ε, υπευλήθη από ε, τη συνάδελφο Τρούπελ. Αλλά παρακαλώ για την προθεσμία, για τις τροπολογίες. Δεν την βλέπω, δεν την άκουσα, δεν την, βλέπω στο έντυπο να σας πω. Γιατί δεν το είπα ακόμα. Το λέω τώρα και στο τέλος θα το ξαναπώ. Και για τις δύο εκθέσεις, και για την έκθεση της κυρίας Τρούπελ και για την έκθεση του κυρίου Τζαμπάτσκι, είναι 26 Ιανουαρίου στις 2 το μεσημέρι. 26 πρώτου 17 στις 2 το μεσημέρι. Λίγη προθεσμία για τις τροπολογίες σας. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τον κύριο Τζαμάνσκι να μας παρουσιάσει τη δική του έκθεση και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η συνθήκη του Μαρακές εγκρίθηκε το 2013 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοτικής Διδιοκτησίας και έχει υπογραφεί από περισσότερες από 60 χώρες συμπεριλαμβανομένης Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κρατών μελών της. Βασικός στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύνολο υποχρεωτικών εξαιρέσεων και περιορισμών για τους τυφλούς, για τα άτομα με μειωμένη όραση και τα άτομα με άλλα προβλήματα ανάγνωση εντύπων. Τώρα οι εξαιρέσει αυτές και περιορισμοί στα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησίας που θα πρέπει να εισαχθούν σε όλα τα υπογράφοντα μέρη θα επιτρέπουν την παραγωγή, τη διανομή και τη διαθεσιμότητα των δημοσιευμένων έργων σε μορφότυπους σχεδιασμένους έτσι ώστε να είναι διαθέσιμοι για τυφλούς, για άτομα με μειωμένη όραση και για άτομα με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων. Και προκειμένου να είναι δυνατή η διασνοριακή ανταλλαγή των εν λόγω έργων. Και ουσιαστικά η ανταλλαγή αυτή είναι ο σκοπός του παρόντος κανονισμού που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ και η πολιτική μου ομάδα πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Στο Συμβούλιο υπήρξε μια κάποια παρανόηση για το ποιος θα πρέπει να επικυρώσει τη συνθήκη αυτή και πότε θα πρέπει να επικυρωθεί. Το αποτέλεσμα του κανονισμού αυτού θα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να συνάδει πλέον με τα όσα λέγονται στη συνθήκη του Μαρακές όσον αφορά τη διασυνοριακή ενταλλαγή έργων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που είναι συμβαλόμενα μέρη στη συνθήκη του Μαρακές είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποιοι είναι οι ορισμοί αυτή τη στιγμή που προτείνονται, ποιο είναι ο δικαιούχο, τι είναι τα αντίγραφα σε προσβάσιμο μορφότυπο και ιδίω ποιε είναι οι οντότητε που έχουν λάβει άδεια διανομή, κοινοποίηση και διάθεση στου ενδιαφερόμενου δικαιούχου των αντιγράφων σε προσβάσιμο μορφότυπο. Επίση, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι οι εξαγωγέ των έργων αυτών δεν θα οδηγήσουν σε εμπορικά προβλήματα και είναι σημαντικό να υπάρχει ασφάλεια δικαίου για τις εξισοδοτημένες οντότητες που είναι κατεστημένες σε κράτος μέλος όταν ασχολούνται με διασυνοριακές δραστηριότητες με τρίτες χώρες. Πιστεύω ότι ο κανονισμός αυτός θα πρέπει μέσω εντός πέντε ετών να αναθεωρηθεί. Και τονίζω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει αυτός ο κανονισμός. Πολλοί συνάδελφοι διάβασαν το σχέδιο αυτό γνωμοδότησης και επίσης τη γνωμοδότηση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών συμφωνούν με τις τροπολογίες μου, με την εξαίρεση της τροπολογίας 4. Και αυτό διότι πιστεύουν ότι η τροπολογία αυτή μειώνει τον αριθμό των εξοδοτημένων φορέων. Τώρα, ο λόγος για τον οποίο επέβαλα την τροπολογία αυτή είναι το ότι αντιστοιχεί στο άρθρο 2 σημείο 6 της συνθήκης του Μαρακές. 2 γάμα με συγχωρείτε. Είναι λογικό θεωρώ να εξειδωτούνται οι φορείς αυτοί από τις αρμόδιες κυβερνήσεις τους. Προφανώς μπορώ να αναθεωρήσω το κείμενο της γνωμοδότησης αυτής, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνωμοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών. Για μια ακόμη φορά, όπως ακούσαμε, η πέμπτη είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών, πέμπτη 26 του μηνός 2 το μεσημέρι. Ευχαριστώ τη Γραμματεία και ευχαριστώ και εσάς για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τζαμάνσκι. Ο Λουίτζι Ευχαριστώ πρόεδρε. Όσοι σκιώδης ε, για το S&D να συμφωνήσω με τα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Θετική ανταπόκριση λοιπόν για την πρόταση οδηγίας και κανονισμού της Ιεραρχικής Επιτροπής. Διότι πρέπει να ευθυγραμμίσουμε το ευρωπαϊκό δίκαιο προς τις ε, διεθνείς δεσμεύσει που έχει αναλάβει η Ένωση. Τα μεγέθη τα θύμισαν οι συνάδελφοι, αλλά πίσω από τα μεγέθη κρύβονται άνθρωποι. Τα δεδομένα του 10 μιλούν για 2,5 εκατομμύρια τυφλούς και 20 και άνω εκατομμύρια άλλους ανθρώπους, άλλους πολίτες με προβλήματα οράσεως, μειωμένης οράσεως δηλαδή εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμα της 3ης Φεβρουαρίου του 2016 έχουμε δεσμευθεί λέγοντας ότι πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία της επικύρωσης της Σύμβασης του Μαρακές για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα υπόλοιπα ελέγξαν ήδη και δεν θα τα επαναλάβω. Τώρα, και η κυρία Τρούπελ και ο κύριος Τζαμπάσκι θύμισαν κάποια ζητήματα τα οποία θα ήθελα να υπογραμμίσω και εγώ. Η πρόταση του κανονισμού συνδέεται άμεσα με την οδηγία, διότι η οδηγία περιγράφει το περιεχόμενο των εξαιρέσεων που θα επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο κανονισμός αναφέρεται στις διασυνοριακές ε, ανταλλαγές και τους μορφοτύπους που θα επιτρέπονται μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τριτών χωρών. Συνυπογραφόντων, δηλαδή, του Μαρακές. Τα δύο πλαίσια είναι παρόμοια. Οι ορισμοί είναι ταυτόσιμοι και αυτό είναι σημαντικό διότι μας επιτρέπει να έχουμε μια συνεκτική προσέγγιση και επομένως θεωρώ ότι οι τροποποιήσεις που έχουν γίνει δεν είναι ε, κρίσιμη ουσιαστική σημασία, αλλά χάρη ασφαλεία δικαίου για όλους τους ενδιαφερομένους φορείς κάποια εδάφια θα πρέπει να διαφημιστούν. Το, έκανε, το έπραξε ήδη ο κύριος ε, Τζαμπάσκι ε, στο σχέδιό του, ευθυγραμμένως περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση στην σύμβαση του Μαρακές και επιφυλασσόμεθα να υποβάλουμε αυτές τις τροπολογίες, σχετικά δηλαδή με αυτό το θέμα, και μία πρόταση, επιτρέψτε μου, που δεν περιέχεται στην πρόταση της Κομισιόν. Δηλαδή, τη δημιουργία μιας τράπεζας δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωσης, ώστε να αποφύγουμε περιτές και επαχθεί έρευνες επί δεδομένων που είναι ήδη διαθέσιμα. Δημιουργώντα ένα ενιαίο database η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με τη βιβλιογραφία των έργων που έχουν παραχθεί σε μορφοτύπους προσβάσιμους ώστε να έχουμε μια ενιαία τράπεζα δεδομένων ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι ε, αυτό το έργο θα μπορούσε να έχει ένα κόστος, αλλά θα μπορούσαμε να αποφύγουμε πολύ σημαντικό άλλο κόστος τυχών διαφορών που θα μπορούσαν να απορρέουν χωρίς να έχουμε ένα πλαίσιο που να εγγυάται τη χρήση των μορφωτύπων αυτών. Προκειμένου να επιτρέψουμε δηλαδή σε όλους από την ε, διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, συμφωνούμε φαντάζομαι όλοι ότι πρέπει να επιτύχουμε την σωστή ισορροπία ώστε να αποφεύγονται αποκλήσεις σχετικά με εκείνο που πρέπει να εγγυηθούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θέλει να τοποθετηθεί. Yeah, Θέλετε, παρακαλώ. lot, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Θα είμαι σύντομος. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ήθελα πρώτα απ' όλα να επαναλάβω ότι η Κοψιόν χαιρετίζει την προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο φάκελο αυτό υπάρχει μια γενική αναγνώριση ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι ισορροπή, πηγαίνει στην σωστή κατεύθυνση και υπάρχει μια γενική συμφωνία που όλοι επιθυμούμε να υπάρχει επαρκής νομοθεσία ώστε να υλοποιηθεί η συνθήκη, η σύμβαση το συντομότερο δυνατόν και το ομαλότερο δυνατόν. Μας ικανοποιεί λοιπόν το γεγονό ότι υπάρχει μια κοινή κατανόηση των στόχων μας. Τώρα, η πρώτη οδηγία και κανονισμού σχετίζονται άμεσα. Αυτό εξηγήθηκε ήδη από τους εισηγητές και από αρκετούς άλλους ομιλητές. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω. Σχετίζονται διότι με την οδηγία καλύπτουμε τα θέματα της εσωτερικής αγοράς ως προς το μηχανισμό, εναρμονίζουμε δηλαδή τις εξαιρέσεις χάρη των τυφλών και ανθρώπων με μειωμένη όραση, ώστε να έχουμε τους ίδιους κανόνες δηλαδή παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να αρμονίζουμε και τις ανταλλαγές μεταξύ των εξιωτημένων αρχών και των δικαιούχων εντός της ιστορικής αγοράς. Με τον κανονισμό καλύπτουμε τις εισαγωγές και εξαγωγές με τρίτες χώρες. Υπάρχει λοιπόν Λόγο και ανάγκη να έχουμε μια κοινή προσέγγιση μεταξύ των δύο αυτών πεδίων με κοινού ορισμού. Δικαιούχου, εξωτημένε αρχέ, ε, εξωτημένου μορφοτύπου κτλ. Ε, κάτι τελευταίο καθότι εθίχθηκε στην συζήτηση των ορισμών. Η προσέγγιση της Κομισιόν είναι να είναι απολύτως πιστή στη συνθήκη δεν θέλαμε άλλες προϋποθέσεις, πρόσθετες προϋποθέσεις ή εξωτερικούς παράγοντες, γιατί θεωρούμε ότι το πνεύμα της συνθήκης μπορεί με αυτόν τον τρόπο να καλυφθεί πιστότερα. Θα έπρεπε να πούμε ότι ως προς κάποιες πτυχές έχουμε μια μικρή απόκληση από την διατύπωση της συνθήκης. Αυτό όμως όχι προκειμένου να έχουμε τροποποίηση επί της ουσίας, αλλά στις περισσότερες ε, περιπτώσεις και κυρίως εδώ μιλούμε για τις εξουσιοδοτημένες αρχές φορείς, προσπαθούμε να απλουστεύσουμε χάρη ασφαλεία δικαίου τον όρο αυτό, την ορολογία, ώστε να προσαρμόζεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Η έννοια του εξουσιοδοτημένου φορέα υπό την έννοια του κανονισμού είναι η ίδια ακόμα και αν διατυπώνεται ελαφρώς διαφορετικά από το άρθρο 2 της συμβάσεως. Δεν πρέπει να υπάρχει λοιπόν κάποια παρανόηση σχετικά με αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή ουσιαστική παρέκκληση. Υπάρχει μια διαφορετική διατύπωση ελαφρώς. Κάτι που είναι σημαντικό να διατηρούμε υπόψη εδώ είναι το θέμα εξουσιοδοτήσεων και του κατά πόσον η σύμβαση απαιτεί από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν συστήματα αξιοδότησης συγκεκριμένα. Η αναφορά στον εξουσιοδοτημένο ή αναγνωρισμένο φορέα δεν σημαίνει υποχρεωτικές εξοδοτήσεις που θα έπρεπε να παρέχουν τα κρατημέλη. Και δεν νομίζω ότι αυτό το εξοδοτημένος ή αναγνωρισμένος που βλέπουμε στη διάταξη θα πρέπει να το ερμηνεύσετε ως προεξουσιοδοτήσεις ή αυτοματοποιημένες εξουσιοδοτήσεις και το βλέπω και στο άρθρο 4 πάφος σε τη σύμβαση του Μαρακέσου όπου παραπέμπουμε σε άλλους φορείς, άλλους οργανισμούς μη κερδοσκοπικούς κτλ. Και σύμφωνα με την δική μας ανάλυση, στα κράτη-μέλη έχουμε πολύ διαφορετικές ε, περιπτώσεις, καταστάσεις. Έχουμε δηλαδή οργανισμούς και φορείς που είναι εξαιρετημένοι για τέτοιου είδους δραστηριότητες, που δεν έχουν προ εξουσιοδότηση, προηγούμενη εξουσιοδότηση κυβερνητική. Προκειμένου λοιπόν να είμαστε πιστοί προς τους στόχους της σύμβασης, ε, πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι όταν μιλούμε για εξουσιοδότηση. Και η προηγούμενη αυτή εξουσιοδότηση ή αδειοδότηση θα μπορούσε να είναι ένα πλαίσιο για κυβερνητικές αρχές να εξαιρέσουν φορείς που διαφορετικά θα ήταν δικαιούχοι είναι κάτι επί του οποίου κατά την άποψη της Κομισιόν πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Όμως, και εδώ η διαφορετική διατύπωση δεν σημαίνει και ουσιαστική απόκληση. Εδώ θα μείνω πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Χέλγα Τρούπελ δεν ξέρω αν θέλει ξανά. Θέλει. Πολύ γενικά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους σε γενικές γραμμές είπαν ότι θέλουν να ακολουθήσουν την πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να μην αλλάξει η πρόταση, αλλά να αλλάξει η κατάσταση για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Ε, περιμένω με ενδιαφέρον τις τροπολογίες για να δούμε τις λεπτομέρειες και πού μπορούμε να βρούμε μια κοινή γραμμή και συμβιβασμό. Αλλά γενικά θα έλεγα και πάλι ότι ας εργαστούμε σε καλό πνεύμα για να βρούμε μια καλή λύση για τους τυφλούς και τους ανθρώπους με προβλήματα όρεσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Τζαμπάσκι, θέλετε να πείτε τίποτα. Όχι, μια χαρά, όλα καλά. Ωραία. Θα ήθελα να σας πω το εξή τώρα. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, Γιούρι, ε, κάνει ακρόαση για τις ημεσουμαρακές στις 30 Ιανουαρίου, 5 ε, με μάλλον στις 3 με 4 το απόγευμα Έχετε λάβει όλοι τις προσκλήσεις, ε, θα το βρείτε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και αν ενδιαφέρεστε είστε προσκεκλημένοι στην ακρόαση αυτή. Επαναλαμβάνω, ε, προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 26 Ιανουαρίου στις 2 το μεσημέρι. Η δε ψηφοφορία θα γίνει στις 28 Φεβρουαρίου εδώ στην Επιτροπή μας. Και θα τα δούμε με την Επιτροπή Γιούρη Δομικών Θεμάτων. Αν 27 το μηνός θα ψηφίσουμε, λάθο Ο κατάλογο μου. 27 του ενό θα ψηφίσουμε και θα το διαπραγματευτούμε με την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να αναβάλουν λίγο τη δική τους ψηφοφορία για να μπορέσει να φτάσει η γνωμοδότησή μας και να ληφθεί υπόψη και στην τελική του ε, έκθεση. Ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή συνεδρίαση. Μου διευκολύνατε πολύ τη ζωή να προεδρεύσω και στις ψηφοφορίες που ήταν και μαραθώνιος. Καλά τα καταφέραμε από κοινού. Δεν θέλω να σας αφήσω να φύγετε για μεσημέρι χωρίς να σας θυμίσω ότι το απόγευμα στις 3 η ώρα έχουμε ακρόαση. Και σας προσκαλώ όλους θερμότατα και θα χαρώ να σας ξαναδώ όλους στις 3 η ώρα για την ακρόαση αυτή. Για να μην αισθανόμαστε εδώ τη μοναξιά της ε, εξουσίας. Και οι περιγνώμονες να έχουν την απαραίτητη ε, προσοχή. Ε, Καλή σας όρεξη. Ευχαριστούμε και τους συγκεκριμένους και τις διερμηνείς. Διερμηνείς, ευχαριστώ την Πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε.